Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε στην ώρα μας, γιατί έχουμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Θα περιμένουμε δύο λεφτά ακόμα και μετά θα ξεκινήσουμε. Voilà. And then I ask you, uh, Θα σας παρακαλέσω, σε περίπτωση που χρειαστεί, να φορέσετε τα ακουστικά σας, γιατί θα μιλήσω γερμανικά. So, sehr Μέλη της Επιτροπής, προσκεκλημένοι, σήμερα έχουμε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε αμέσως τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε σήμερα στο πρόγραμμά μας την ε, ακρόαση, μια συναρπαστική ακρόαση, και γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα το χρόνο μα. Στην Επιτροπή μα ξεκινάμε με την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, θεωρούμε ότι είναι εγκεκριμένη. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στι ανακοινώσει τη Προέδρου. Στην συνεδρία τη 6 Νοεμβρίου 2019, οι συντονιστέ αποφάσισαν να ε, αναθέσουν τις εξής εκθέσεις στις εξή στις εξής ομάδες η κάλυψη του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και η συμμετοχή των γυναικών στην ε, ψηφιακή οικονομία στο ΕΛΚ αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την υγεία των γυναικών και πώς έχουν τα πράγματα σήμερα στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η υποστήριξη της ισότητας των ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα των μαθηματικών, της πληροφορικής, των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, MINT, για τους ΡΙΝΙΟΥ η, η των ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο τη εξωτερική πολιτική και τη πολιτική ασφαλείας Ευρωπαϊκή Ένωση στου Πρασίνου. Οι επιπτώσει τη ενδοοικογενειακή βία και τη επιμέλεια των παιδιών ε, για τι γυναίκε στην ΚΟΕ η παρακολούθηση, η έκθεση monitoring για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΚΟΕ και μια έκθεση πρωτοβουλία με τον τίτλο Καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών, βία στο διαδίκτυο, στο ΕΛΚ. Και η έκθεση για την εφαρμογή τη οδηγία για την καταπολέμηση τη ε, εμπορία ανθρώπων στου ΡΙΝΙΟΥ. Η δήλωση για την διακριτική μεταχείριση εξαιτία του ε, στα διάφορα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και το Φόρουμ τη Ισότητα των ε, Γενεών στο πλαίσιο τη ερχόμενη ε, συνεδρίαση είναι κάτι που θα το οργανώσουμε, καθώ και ένα ταξίδι στο Μεξικό το Μάιο του 2020 για το Generation Equality Forum. Μετά περνάμε στο 2-2. Η συμμετοχή μιας γυναι... ομάδας γυναικών από την Κένια που ήταν φιναλίστ στο show Mrs. President ε, στην Κένια. Είναι σήμερα προσκεκλημένες και μαζί μας στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι θα έχετε όλοι την ευκαιρία να πάρετε μέρο σε ένα κοκτέιλ. Σήμερα δεν θα έχουμε χρόνο για παρεμβάσει ή τοποθετήσει προφορικέ, γιατί έχουμε πολύ φορτωμένη μέρη σε διάταξη. Αλλά εκεί θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τι υποψήφιέ μα, τι φιναλίστ. Και είχα την ευκαιρία να τι γνωρίσω εγώ προσωπικά προηγουμένω. Και θα ήθελα απλώ σήμερα να πω ότι θα δώσω λόγο, το λόγο μόνο στην νικήτρια του σοου, την κυρία Νερία Οκέτς. Ε, εάν μπορείτε να μας πείτε πολύ λίγα λόγια για το ποια είστε, να συστηθείτε και να μας πείτε γιατί αποφασίσατε να, να συμμετέχετε σε αυτό το show, τι στόχο είχε, γιατί ξέρουμε ότι ήταν ε, πολύ επιτυχημένο και καινοτόμο και έδειξε τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στην Κένια και να τις υποστηρίξει. Ίσως μελλοντικά να υπάρξουν όντως κυρίες πρόεδροι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Είναι τιμή μου για τις φιναλίστες και για μένα να είμαι εδώ σήμερα στην Επιτροπή αυτή. Για τις γυναίκες ε, της Κένιας χαιρόμαστε που έχουμε τη δυνατότητα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουμε το ταλέντο μας ε, στο να ηγηθούμε σε όλο τον κόσμο. Το Κοινοβούλιο στη χώρα μας δεν έχει όμως νομοθετήσει έτσι ώστε κάθε θεσμικό όργανο και το Κοινοβούλιο να έχει ισότιμη εκπροσώπηση. Πολύ συχνά ρωτάνε όλοι τι πρέπει τελικά να κάνουν οι γυναίκες. Γιατί δεν μπορούν να δώσουν μια μάχη για την ηγεσία της χώρας τους όπως οι άντρες. Είναι πλέον ε, μια πραγματικότητα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουν οι Κενιάτες τι προσφέρουν οι γυναίκες πριν από τις εκλογές. Και όσο πλησιάζουμε προς το 2022 είναι πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα να δημιουργήσει μια ορατότητα συνεχή, όχι μόνο για τις πέντε, ε, εμάς τις πέντε, αλλά για όλες τις άλλες γυναίκες οι οποίες δίνουν, οι οποίες δίνουν αυτή τη μάχη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι μια γυναίκα που έχει φωνή στο σπίτι της δεν θα εξασφαλίσει μόνο την υγεία για τα παιδιά της και τα, παιδιά της Κένιας θα τα προγραμματίσει αυτά η κυβέρνηση ε, θα εξασφαλίσει υγεία θα σκεφτεί μια γυναίκα στην ε, ε εξουσία ότι θα πρέπει να δοθούν χρήματα για την εκπαίδευση των παιδιών γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή τη φωνή εγώ και οι υπόλοιπε φιναλίστες έχουμε πλέον μια πλατφόρμα για να διαπραγματευτούμε έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από όλα τα κόμματα ότι πλέον εμείς οριμάσαμε και θα δώσουμε τη μάχη για, αυτές τις, για αυτά τα αξιώματα. Ε, θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει ορατά αυτές τις γυναίκες που θέλουν να ε, παρουσιαστούν στις εκλογές το 2022. Θέλουμε να υπάρξει στήριξη, για να έχουμε project που να έχουν σχέση με τις κοινότητές μας. Το θέμα, παραδείγματος χάρη, των ε, γυναικών, ε, των κοριτσιών που είναι έγκυες σε πολύ μικρή ηλικία. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η υποστήριξή σας. Είναι επίσης σημαντικό Εμείς υποστηρίζουμε, ε, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δημιουργηθεί, δημιουργήσει αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει αυτή η χρηματοδότηση όντως να πάει σε γυναίκες που μπορούν να προωθήσουν κάποια ζητήματα και να υπάρχει μια εταιρική σχέση η οποία να είναι μακροπρόθεσμη. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να μας δώσετε για την ισότητα των άντρων και γυναικών στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όπως είπατε, Ελπίζουμε και εμείς ότι θα μπορέσουμε στη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής να ε, επωφεληθούμε και εμείς από την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε και να το χρησιμοποιήσουμε επικοδομητικά και στο δικό μας μέλλον. Ε, μέλλον. Ε, περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μέσα διάταξης για την ε, οργάνωση της ακρόασης για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Ήθελα να καλέσω και να, πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω όλους τους ε, προσκεκλημένους μας και κυρίως να καλέσω τις εμπειρογνώμονές μας που είχαν την ε, ευγένεια να είναι εδώ σήμερα μαζί μας να έρθουν εδώ για να ε, ξεκινήσει η ακρόαση με θέμα την ημέρα αυτή για την καταπολέμηση, την εξάλληψη της βίας των γυναικών. Ε, μια ημέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου και είναι μια ευκαιρία να έχουμε μια επισκόπηση για το τι έχει συμβεί σε διεθνές επίπεδο για το θέμα αυτό και τι μέτρα έχουν αναλυφθεί. Τα στοιχεία που έχουμε πραγματικά μας ε, κάνουν να ανησυχούμε και γιατί συγκεκριμένα μία στις τρεις γυναίκες ή κορίτσια έχουν υποφέρει στη διάρκεια της ζωής τους από σωματική σεξουαλική βία και συνήθως από τον ίδιο του τον σύντροφο, τα μέλη τη οικογένεια του από, το άμεσο, από τον άμεσο περίγυρό τους. Το 52% των ύπανδρων ε, ε, όσων βρίσκονται σε μία σχέση μόνιμη, πολλές, σπάνια έχουν, δεν μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα για τη σεξουαλική επαφή ή τα μέτρα αντισύλληψη ή την ε, προστασία τη υγεία του. Επίση, διεθνώ 790 εκατομμύρια γυναίκε ή κορίτσια έχουν παντρευτεί πριν το 18ο έτος τη ηλικία του. Δηλαδή, μιλάμε για το kinder child marriages, όπω λέγεται, τους γάμου παιδιών, καταναγκαστικού γάμου, που είναι σήμερα ένα πολύ επίκαιρο θέμα εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια είναι ε, όπως και παλιότερα ε, θύματα του ε, γυναικείου ακροτηριασμού των γυναικείων του εκτοτηριασμού μάλλον των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της κλειτοριδεκτομής. Μία στις δύο γυναίκες το 2012 που είχε χάσει τη ζωή του είχε δολοφονηθεί από μέλος της οικογένειάς της ή το σύντροφό τη, Αυτά είναι στοιχεία που πραγματικά πρέπει όλοι να τα δούμε με μεγάλη προσοχή και θα πρέπει να κοιτάξουμε να βελτιωθούν τα όσα συμβαίνουν. Ε, το 71% των θυμάτων ε, της εμπορίας ανθρώπου είναι, ανθρώπων είναι γυναίκες ή κορίτσια. τρεις από τέσσερις ε, από τις γυναίκες αυτές οι κορίτσια έχουν μάλιστα πέσει και θέμα σεξουαλικής βίας. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια της Διεθνούς ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να δούμε τι συμβαίνει με την κατάσταση αυτή στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώ έχουν λάβει μέτρα για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών με σχετικέ διαδικασίε. Θα πρέπει να έχουμε μια ανταλλαγή απόψε για το θέμα αυτό. Η ακρόαση αυτή έχει οργανωθεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα της δημόσιας ακρόασης προβλέπει να ε, δούμε με τις εμπειρογνώμονές μας, ε, τις προσκεκλημένες μας, ε, μια επισκόπηση, μια συνοπτική εικόνα για το ποια είναι τα διεθνή μέτρα, ένδικα μέσα που προσφέρονται για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε τα συγκεκριμένα μέτρα των κρατών μελών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Και θα δούμε και έναν οδηγό της ΕΓΕ, του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, που δημιουργήθηκε για την ε, υποστήριξη των αστυνομικών αρχών σε σχέση με το θέμα αυτό. Θα πρέπει επίσης να σας παρακαλέσω να προσπαθήσουμε όλοι να σεβαστούμε το χρόνο ε, ομιλίας. Ε, δέκα λεπτά για την κάθε προσκεκλημένη μας λοιπόν το πολύ και μετά θα έχουμε και την ευκαιρία για ένα γύρο ερωταπαντήσεων. διότι θα πρέπει να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε γέρο την ακρόασή μα. Εάν δεν σεβαστούμε τα όρια, δεν θα είναι αυτό εφικτό. Θα ήθελα λοιπόν απευθεία να δώσω το λόγο στην πρώτη από τι προσκεκλημένε μα, που θα μα μιλήσει για τα διεθνή ενδικά μέσα, η οποία είναι η κυρία Μασλίν, Μασλίν Ναουντή. Με συγχωρείτε, προσπαθώ να μην κατακριοργήσω τα ονόματά σας, δείξετε κάποια κατανόηση. Θα μας μιλήσετε για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών σε, και την ενδοοικογενειακή βία και το τι γίνεται με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τα διδάγματα που αντλήσαμε από την παρακολούθηση χωρών από την οργάνωση Γκρέβιο. Κυρία Νάουντι, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, κύρια Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την πρόσκλησή σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα ως πρόεδρος του Γκρεβιό να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτήν την ακρόαση. Και όπως όλοι γνωρίζετε, η ομάδα μας στο Γκρέβιο είναι η ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω για τα πορίσματα της παρακολούθησης μας και μετά να δούμε κάποιες από τις τάσεις που έχουμε παρατηρήσει αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ισχύει εδώ και πέντε χρόνια, έχει επικυρωθεί από 34 κράτη μέχρι στιγμής και έχει υπογραφεί από 11 ακόμη, καθώς επίσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μπορεί να επικυρωθεί και από χώρες που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουμε μία χώρα προκειμένου την, την Ισία η οποία έχει α, συμμετάσχει και αυτή. Είναι καλό να βλέπουμε ότι επεκτηνόμαστε και πέρα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι ευρέως αποδεκτή στην σκηνή των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι εξαιρετικά καινοτόμο και βεβαίως χάρη στην δική μας ομάδα έχει εμπνεύσει πολλές σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία αλλά και στην πρακτική η ομάδα μας, η ομάδα παρακολούθησης κάθε χώρας καταλήγει και σε μία συγκεκριμένη αναφορά της νομοθεσίας που ισχύει σε τοπικό επίπεδο. Και τώρα που έχουμε ολοκληρώσει αρκετές από αυτές τις αξιολογήσεις, μας έχει δώσει και μία γενική εικόνα των βέλτιστων πρακτικών, καθώς επίσης και των προκλήσεων που έχουμε εντοπίσει όταν ε, κοιτάζουμε λοιπόν τις αναδυόμενες τάσεις αλλά και τις προκλήσεις μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία αυτή παρακολούθησης είναι κάτι θετικό. Η ομάδα μας κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων και των εκθέσεων που συντάσσουμε έχει εντοπίσει καλή θέληση από τις ε, κυβερνήσεις. Δουλεύουμε σκληρά για να εξασφαλίσουμε το ότι έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο μέσω της παρακολούθησης που κάνουμε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή όχι μόνο με τις κυβερνήσεις αλλά και με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Και μέχρι στιγμή το feedback που έχουμε λάβει, καθώς και τα σχόλια των κυβερνήσεων σε σχέση με τις διάφορες εκθέσεις μας, τις οποίες στέλνουμε στη χώρα αφού τις ολοκληρώσουμε και οι κυβερνήσεις μπορούν με τη σειρά τους να μας δώσουν και αυτοί τα δικά τους σχόλια. Και αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να χτίσουμε εμπιστοσύνη με τα διάφορα κράτη-μέλη. Και σε γενικές γραμμές οι κυβερνήσεις των κρατών αποδέχονται τις συστάσεις που κάνουμε στις εκθέσεις μας. Επίσης, είμαστε αρκετά τυχεροί και καλωσορίζουμε την ευκαιρία που είχαμε πρόσφατα στην Φινλανδία και γιατί το αναφέρω αυτό ως μια βέλτιστη πρακτική αλλά και σαν έμπνευση. Αυτό είναι μια καλή ιδέα. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς ίσως να σκεφτεί κάποιος. Μας προσκάλεσαν και πάλι πίσω στη χώρα, μέσως μετά την έκδοση της έκθεσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε επιπλέον με τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό βοηθάει να αυξηθεί η ορατότητα της έκθεσης που συντάξαμε και μας ε, βοηθάει επίσης τόσο τις αρχές όσο και τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, τους δίνει μια καλύτερη ιδέα του πώς να προχωρήσουν από τη συστάση μας και μετά. Ενθαρρύνω λοιπόν τα, τα κράτη που πολύ σύντομα θα περάσουν από αξιολόγηση να σκεφτούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, μέσω της διάφορες α, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με κυβερνητικών οργανισμών, κυβερνήσεις κτλ. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε εκδώσει εννέα εκθέσεις με μία δέκατη να εκκρεμεί για την Γαλλία, η οποία εκδίδεται σήμερα τα μεσάνυχτα. Είμαστε λίγο σαν τη σταχτομπούτα εδώ. Είναι τρεις ακόμη εκθέσεις οι οποίες αφορούν τρεις άλλες χώρες, έχουν γίνει επισκέψεις σε διάφορες χώρες και έχουμε λάβει και τοπικές εκθέσεις και από άλλα εμπλεκόμενα μέρη σε διάφορα κράτη, που σημαίνει ότι περίπου μισά από τα κράτη που συμμετέχουν στην σύμβαση είναι ήδη ενεργά σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης. Τι έχει αλλάξει λοιπόν ως αποτέλεσμα τόσο της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης όσο και της συνεχούς παρακολούθησης. Λοιπόν, χάρη στη σύμβαση αρκετοί νόμοι έχουν αλλάξει. Νέα εργαλεία υπάρχουν, πολιτικές έχουν αναθεωρηθεί σε διάφορες χώρες. Να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα η υιοθέτηση νομοθεσιών που καθορίζει τη σεξουαλική παρενόχληση και την ε, παρακολούθηση, κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι στιγμής, ο ορισμός της έλλειψης συγκατάθεσης, η οργάνωση διαφόρων επιτροπών μεταξύ ε, διάφορων φορέων, κάτι το οποίο έγινε στην Αλβανία. helplines, 24... Ο ορισμός του βιασμού η συγκρότηση τηλεφωνικών γραμμών, κάτι το οποίο έχει, έχουμε δει στη Γερμανία, η δημιουργία καταφυγίων, δημόσιων καταφυγίων στο Μαυροβούνιο, η εισαγωγή της βίας εναντίον των γυναικών ως ακαδημαϊκό αντικείμενο ή ενημέρωση, εκπαίδευση νομικών εμπειρογνωμόνων, όπως για παράδειγμα στη Σουηδία, η ειδική εκπαίδευση για εισαγγελείς, για δικηγόρους στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όλες αυτές είναι θετικές εξελίξεις. Κάποιες χώρες ήδη είχαν εφαρμόσει τέτοιου τύπου μέτρα, δηλαδή είχαν επικυρώσει τη σύμβαση, άλλες μετά την αξιολόγηση, σε γενικές γραμμές όμως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλες αυτές οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα. Έχουν προκύψει και κάποια ζητήματα, τα οποία βλέπουμε αρκετά συχνά και μπορούμε να, να τα ορίσουμε ως κοινέ προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα, η γενική ικανότητα του να υπάρξουν συγκεκριμένες δομές οι οποίες ακόμη και αν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει μια καταλήλη αρχή, δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και τόσο τα οικονομικά μέσα όσο και οι αρχές είναι πολύ σημαντικές ούτως ώστε να μπορέσουμε να, να έχουμε αυτές τις λειτουργικές δομές. Η συλλογή δεδομένων, η προϋπόθεση συλλογής δεδομένων έχει ενθαρρύνει αρκετές ε, χώρες να μπορέσουν να συγκεντρώνουν στοιχεία σε ό,τι αφορά τη βία εναντίον των γυναικών, τη σχέση μεταξύ των ε, διαφορών ατόμων που διαπράττουν βίες ε, ενέργειες και του φίλου του θύματος. Σε πολλές περιπτώσεις όμως η συλλογή δεδομένων δεν γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες. Είναι πολύ σημαντικό. Τα συστήματα συλλογής δεδομένων δε σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν από τομέα σε τομέα. Δηλαδή από τη μία μεριά έχουμε για παράδειγμα τη συλλογή δεδομένων τη αστυνομία και από την άλλη την ε, συλλογή δεδομένων υγειονομικών υπηρεσιών. Και ω αποτέλεσμα δεν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα. Είναι ε, μικρά-μικρά κομμάτια, τα οποία είναι, κομμάτια τα οποία είναι δύσκολο να τα συνθέσουμε για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Με συγχωρείτε. Σε ό,τι αφορά την προστασία τώρα, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα δυνατότητα του να έχει ένα θύμα την ε, δυνατότητα να λάβει μια εντολή που απαγορεύει το δράστη να το πλησιάσει. Σε πολλές περιπτώσεις όμως δεν γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να βρουν νέους τρόπους αντιμετώπισης και προστασίας των θυμάτων. Επίσης, δυστυχώς, πολύ συχνά υπάρχουν και εξαιρέσεις ό,τι αφορά αυτά τα μέτρα προστασίας, όπου σε πολλές περιπτώσεις ο δράστης και το θύμα έχουν από κοινού την κυδαιμονία ενός παιδιού. Όταν υπάρχουν ζητήματα κυδαιμονίας που λαμβάνονται υπόψη, χωρί να, να, λαμβάνει το δικαστήριο υπόψη του αυτά τα μέτρα προστασίας που μπορεί να είναι ενισχύει. Μπορεί να μην τα γνωρίζουν, μπορεί να μην έχουν ελέγξει, κατά πόσο ισχύει, βρίσκεται ενισχύει ή όχι, ε, μία εντολή προστασίας. Και πάλι σε ό,τι αφορά τις ομάδες στήριξης γυναικών που έχουν πέσει θύμα αδείας, έχουμε δει πρόοδο, αλλά και πάλι είναι αυτό το ζήτημα των οικονομικών μέσων. Σε λίγες περιπτώσεις υπάρχει ένα μακρό πρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης τέτοιου τύπου ε, δομών. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν και όχι ίσως απαραίτητα συνδεδεμένο με τη δική μας ομάδα monitoring, έχουμε αρκετά ανησυχητικά σημάδια σε ό,τι αφορά την κάποια οπισθοδρόμηση που μπορεί να υπάρξει σε ό,τι αφορά το ζήτημα προστασίας των γυναικείων δικαιωμάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά τα θύματα βίας και σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγική υγεία, αλλά και την ιδεολογία που έχει να κάνει με την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. κυρίως σε ό,τι αφορά παρερμηνίες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν χώρες που καθυστερούν να επικυρώσουν τη σύμβαση. Ένα χρόνο πριν, μίλησα α, με, κάποιους, με κάποια άτομα σε κάποια από αυτές τις χώρες που ε, με κατηγόρησαν ότι πήγα, εκεί για να τους, ότι πήγα εκεί για να τους κλέψω τα παιδιά. Η απάντησή μου ήταν ότι μου αρέσουν τα παιδιά, αλλά δεν ήρθα εδώ για να κλέψω τα δικά σας. Αυτό όμως είναι το επίπεδο παρερμηνίας που πολλές φορές πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε παθητικοί απέναντι σε, αυτό, σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα και μπορεί να γνωρίζετε και τα ερωτήματα και τα πορίσματα της Επιτροπής της Βενετίας. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα της, Ερμηνεία, της Αρμενίας, με συγχωρείτε, αλλά σε γενικές περιπτώσεις, αυτό που, σε γενικές αυτούς προσπάθησαν να κάνουν ήταν να διασαφηνίσουν κάποιες ε, τέτοιου τύπου παρερμηνίες ή παραπληροφόρηση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εξέλιξη. Όμως θα πρέπει τα κράτη που έχουν επωφεληθεί ως μέλη της σύμβασης ή που έχουν αξιολογηθεί από την ομάδα μας να είναι πιο ενεργά σε ό,τι αφορά τη στήριξη της σύμβασης και να μας δείξουν με αποτελέσματα περί τίνος πρόκειται, ποιες είναι οι πραγματικές αλλαγές δηλαδή που έχουν επιτευχθεί. Χρειαζόμαστε πιο ισχυρή, πιο ενεργή πολιτική δέσμευση από τις κυβερνήσεις οι οποίες στηρίζουν το σκοπό μας. Είναι ανάγκη να δίνουμε πάντοτε το καλό παράδειγμα. Πρέπει να δείχνουμε ότι η βία εναντίον των γυναικών αλλά και όλη η προσπάθειά μας εξάλληψης της βίας εναντίον των γυναικών δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από μια σαφή ιδέα της Ευρώπης. Είναι κάτι, το οποίο, είναι κάτι για το οποίο παλεύουν οι γυναίκες σε όλες τις χώρες. Μπορώ να έχω 1,5 λεπτό ακόμα, λέει ο μιλήτρια. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακόμα και αν με σταματήσετε τώρα, Έχω ολοκληρώσει τη σκέψη μου. Αν μου επιτρέπετε λίγο παραπάνω χρόνο όμως ακόμη, η ομάδα μας κοιτάζει και προς το μέλλον δίνουμε τους αγώνες που πρέπει να δώσουμε, κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, αλλά κοιτάζουμε και προς το μέλλον πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άλλου τύπου ανησυχητικές τάσεις ή να έχουμε και νέες γραμμές δράσης. Πρόσφατα λοιπόν είχαμε ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κοιτάζουμε την δυνατότητα να μπορούμε να προετοιμάσουμε παρεμβάσεις στο δικαστήριο για περιπτώσεις που αφορούν ε, υποθέσεις βίας εναντίον των γυναικών. Επίσης, εξετάζουμε το ζήτημα της βίας στον κυβερνοχώρο. Και το κατά πόσο γνωρίζουμε το τι συμβαίνει, κατά πόσο μπορούμε να αναλάβουμε δράση, όλα αυτά είναι τάσεις που διαρκώς κερδίζουν momentum. Προσπαθούμε να συλλέγουμε στοιχεία, ούτω ώστε και εμείς να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη άποψη πάνω στο ζήτημα αυτό. Και επίσης τα χρόνια περνούν και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε να κοιτάζουμε την εφαρμογή των συστάσεων στις πρώτες χώρες που έχουμε ήδη αξιολογήσει η ομάδα μας στην και ποιες θα είναι οι α, προτεραιότητες του δεύτερου κύματος αξιολογήσεων. Και πάλι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας αυτήν εδώ την ακρόαση και για την προσοχή σας. Ελπίζω ότι δεν θα είναι ένα και μοναδικό γεγονός. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα εξακολουθήσει γιατί πιστεύω ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πολύ. So, herzlichen Dank. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ναουδή. Και τώρα θα προχωρήσουμε αμέσω στη Γενική Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, Τζοάννα Μέικοκ. Καλώ ήρθατε, έχετε το λόγο. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και την Επιτροπή Γυναικών που με προσκάλεσε εδώ σήμερα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τους νέους ευρωβουλευτές αλλά και τους παλαιότερους για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας, για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών εκπροσωπεί χιλιάδες οργανώσεις γυναικών στην Ευρώπη. Ε, θέλουμε να συνεργαστούμε λοιπόν με την Επιτροπή Γυναικών για να προωθήσουμε τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών και να βάλουμε τέλος στην βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Το η οργάνωσή μα ε, συνεργάζεται με τα μέλη μα ανά την Ευρώπη και με τα ευρωπαϊκά όργανα τη Ένωση, ζητώντα ε, να ληφθεί υπόψη σοβαρά η βία κατά των γυναικών και να αποτελέσει προτεραιότητα για να δημιουργήσουμε την κοινωνία που θέλουμε. Όχι να μειώσουμε τη βία, να την εξαλείψουμε. Να την εξαλείψουμε παντελώ. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη όταν οι γυναίκε φοβούνται για την ασφάλειά του στο σπίτι του, στο χώρο εργασία του, στου δημόσιου χώρου στην Ευρώπη. Υπάρχουμε εδώ και 23 χρόνια. Το παρατήρητο το για την βία κατά των γυναικών έχει δώσει ένα χώρο ακτιβισ... φεμινισμού σε, ακτιβισμού, σε ακτιβιστές, επαγγελματίες, οργανώσεις να ανταλλάξουν πραγματογνωμοσύνη, εμπειρίες ε, να δούμε πού έχουμε προχωρήσει, πού έχουμε πιστοχωρήσει και εκεί προωθούμε την καμπάνια μας, την εκστρατεία μας σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της σύμβασης του, του Ισταμπούλ μεταξύ άλλων. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι στο πάνελ αυτό με εξαιρετικού συναδελφούς εδώ αριστερά μου και οι δύο ε, έχουν συνεργαστεί μαζί μας ε, στα πλαίσια του παρατηρητηρίου ε, της βίας κατά των γυναικών. Έχω 10 λεπτά στη διάθεσή μου, είναι λίγο χρονικό διάστημα διότι πολλά θα ήθελα να πω. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο για να υπάρξει χρόνος και για ανταλλαγή απόψεων, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Να πω δύο λόγια ε, για την ε, βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών ε, πρώτα. Να σας πω ποια είναι η δική μας προοπτική σε ό,τι αφορά το θετικό αντίκτυπο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης επί τόπου από πλευρά δηλαδή από το πρίσμα των οργανώσεων γυναικών, αυτό ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό με αυτό που μόλι ανέφερε η κυρία Νάουντι. Επίση, θα αναφερθούμε σε κάποιε από τι σκέψει μα ε, για τα κενά στην εφαρμογή και βεβαίω τι προκλήσει που έχουμε μπροστά μα και να πω και κάποια πράγματα για το τι περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία ε, για να υποστηρίξει ε, την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Κυρία Πρόεδρε, ήδη αναφερθήκατε ε, στην αύξηση τη γυναίκα κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι παρότι, παρότι έχουμε δεκαετίε πρόοδου σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, έχει σταματήσει αυτή η πρόοδο. Ε, σε καμία χώρα τη Ένωση ή ισότητα μεταξύ ανδρών κόσμο δεν έχει επιτευχθεί ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στην Ευρώπη όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ελεύθερα από την απειλή της βίας ή από την ίδια τη βία. Δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας της ζωής μιας γυναίκας, ενό κοριτσιού, όπου δεν εκτίθεται στη βία και όλες οι μορφές βίας κατά των ανδρών και των κοριτσιών και των γυναικών έχουν τον ίδιο σκοπό. Να κάνουν τις γυναίκες να σιωπήσουν, να μην τους δώσουν την θέση που τους αναλογεί στην κοινωνία. Παίρνει πολλές μορφές αυτή η βία. Υπάρχει ενδοκρινιακή βία, σεξουαλική βία, υπάρχει η παραβίαση σεξουαλικών δικαιωμάτων των γυναικών. Οι γυναίκε και τα κορίτσια, παραδείγματο χάρη, συχνά είναι παγιδευμένε σε συστήματα εμπορία, σε, σε κυκλώματα εμπορία, σε κυκλώματα πορνεία, ε, καθημερινή παρενόχληση στο δρόμο, κύβερνο, βία στον κυβερνοχώρο. Ε, μία στι τρει γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 62 εκατομμύρια γυναίκε δηλαδή, έχουν ζήσει ε, σεξουαλική βία, έχουν ε, την εμπειρία σεξουαλική ε, βία ή βία κατά του σώματό του από την ηλικία των 16 και, μετά. Και βεβαίω ε, παρενόχληση μία στι δύο γυναίκε. Ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 50 γυναίκε πεθαίνουν κάθε εβδομάδα δολοφονημένε από τον σύντροφό του ή από τον πρώην σύντροφό του. Πρόκειται για μια κοινιακοκτονία και πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό οι οργανώσει γυναικών, οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών είναι στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών για δεκαετίες. Έχουμε φέρει αντίγραφα ενός κειμένου που έχουμε προετοιμάσει όπου λέμε πώς θα σταματήσει αυτή η συνεχής βία κατά των γυναικών. Εκεί υπάρχει η ανάλυση μα και οι συστάσει μα για δράσει. Εμεί αναζητούμε λύσει. Πώ μπορούμε δηλαδή να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη όπου οι γυναίκε και, τα κορίτσια δεν θα υπόκεινται στη βία. Έχουμε αφήσει σχετικά αντίγραφα αυτού του εγγράφου ε, εδώ στην αίθουσα, υπάρχει στην σελίδα μα. Ε, και βεβαίω μεγάλη προτεραιότητα για μα είναι να ζητήσουμε την πλήρη εφαρμογή τη σύμβαση τη ε, Κωνσταντινούπολη. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχουν ήδη υποθεί από την κυρία Νάουντι, αλλά πραγματικά συμμεριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό την ανάλυση τη. Η συνθήκη αυτή είναι πολύ σημαντική. Είναι η πρώτη συνθήκη στην Ευρώπη που ποινικοποιεί πολλαπλέ μορφέ βία κατά των γυναικών. Αναγνωρίζει ότι η βία κατά των γυναικών είναι, ανθρώπινο, είναι, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι διάκριση κατά των γυναικών και είναι και αιτίο και αιτιατό τη ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, οι οργανώσεις γυναικών, και εδώ θέλω να το τονίσω, έχουν εργαστεί εντατικά ζητώντας μια τέτοια σύμβαση και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε με πάθος για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης, την επικύρωσή της, για να εξασφαλίσουμε ότι θα τεθεί σε ισχύ ε, για να, για να κάνει πραγματικά τη διαφορά στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε μια χαρτογράφηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη σύμβαση τη ε, Κωνσταντινούπολη μέσα στο παρατηρητήριο μα. Δεν έχουμε ακόμα τελικά αποτελέσματα αυτή τη χαρτογράφηση. Να σα πω κάποια πρώτα στοιχεία όμω. Αυτό που διαπιστώσαμε, το πιο θετικό σε επίπεδο εφαρμογή ε, τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, ε, είναι αυτά που τα οποία έφερε η κυρία Νάουντι ήδη. Σε νομοθετικό επίπεδο, αλλαγέ στην νομοθεσία, αλλαγέ στι πολιτικέ, σε ό,τι αφορά τη διακράτηση των γυναικών. Οι εμπειρογνώμονέ μα έχουν εντοπίσει θετικέ αλλαγέ στου τομεί αυτού σε 17 από τι 23 χώρε. Ε, τι έχουμε αναλύσει. Από τι 17-23 χώρε που αναλύσαμε, μάλλον. Και αυτό είναι θετικό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ε, Βεβαίω, ε, όταν αυτό αποτελεί μέρο ενό ε, εθνικού σχεδίου δράση ή μια εθνική στρατηγική δράση για την καταπολέμηση τη βία, είναι πιο αποτελεσματική η νομοθεσία. Υπάρχουν σειρά παραδείγματα. Ήθελα να μιλήσω και για το βιασμό, αλλά νομίζω αναφέρθηκε ήδη αυτό από την κυρία Νάουντι. Υπάρχει η νομοθεσία ε, για τις σεξουαλικές επιθέσεις 2017 στην Ιρλανδία από την, υπό, Φιτζέρελτ Francis Fitzgerald που είναι και μέλος της Επιτροπής αυτής για που, εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τη σύμβαση της Ισταμπούλ ε, γίνεται αναφορά στη συνένεση για πρώτη φορά σε ένα κείμενο, στη νομοθεσία αυτή συγγνώμη. Επίσης αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως η παιδική πορνογραφία, ε, το grooming, η ποινικοποίηση των ε, υπηρεσιών πορνείας καθώς και η ενδοκρινιακή βία ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι το θέμα της ε, ε κυδαιμονίας των παιδιών. Υπάρχει το θέμα της έλλειψης απαντήσεων στις υπηρεσίες που να ε, λαμβάνουν υπόψη το φύλλο και αυτό έχει επιδεινωθεί βεβαίως ε, λόγω της λιτότητας. Γενικά υπάρχουν τεράστιες περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα στις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ε, όταν μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών, τα δύο τρίτα όλων των καταφυγίων, των καταλημάτων ε, που υπήρχαν για γυναίκες ε, που, είχαν, ε, που έχουν υποστεί ενδοκινιακή βία έχουν κλείσει ή κινδεύουν να κλείνουν στη Ρουμανία. Υπήρχαν γραμμές τηλεφωνικές που μπορεί κάποιος μπορεί μια γυναίκα να τηλεφωνήσει και έχουν πλέον δοθεί αυτές οι γραμμές σε ανθρώπους που δεν έχουν εξειδίκευση, δεν έχουν εμπειρία για τα ζητήματα αυτά ε, της ενδοικογενειακής βίας και βεβαίως ε, αλλού ε, δεν γίνεται τίποτα για τη βία κατά των γυναικών διότι δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία. Η μη επικύρωση επίσης ε, είναι και αυτό ένα ζήτημα και αυτό θα το συζητηθεί και στο επόμενο πάνελ. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι έχουμε και κάποιες προσδοκίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Την ερχόμενη Δευτέρα, όπω είπα, είναι η Διεθνή ημέρα για την κατάργηση τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Οι γυναίκε και τα κορίτσια ανά την Ευρώπη θα βγουν στον δρόμο, θα είμαστε μεταξύ αυτών και τα μέλη μα θα ε, κατέβουν στον δρόμο και στο διαδίκτυο και θα ζητήσουμε. Ε, έχουμε δικαίωμα σε μια ζωή ελεύθερη από βία και από το φόβο τη βία. Θα υπάρξουν πολλέ δηλώσει καλών προθέσεων από του πολιτικού ηθήνοντε ανά την Ευρώπη, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά τα λόγια δεν φτάνουν. Εμείς ζητούμε δράση. Οι, οι φωνές των γυναικών δεν μπορούν να γνωριστούν πια. Είναι πολλές και ακούγονται δυνατά και είμαστε ενωμένε. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε και να ζητάμε για δράση. Πρέπει να λάβουν τι ευθύνε του ε, οι ευρωπαϊκέ αρχέ, έτσι ώστε οι γυναίκε να μπορούν να είναι ασφαλεί και να μην υπόκεινται σε βία. Ε, με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει αναλάβει με μια γυναίκα πρόεδρο, που κατέστησε σαφέ ότι το, η επάλυψη τη βία κάτω των γυναικών προτεραιότητα, για αυτήν ε, έχουμε θαρρυνθεί. Ε, και από το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που είναι εδώ τόσα μέλη σήμερα καταρχήν στην ακρόαση, πολύ, πολλά περισσότερα από ότι στην περσινή ακρόαση. Πραγματικά νιώθουμε ότι αυτό είναι κάτι που μα ενθαρρύνει. Το πρώτο που θα πρέπει όμω να κάνουμε τώρα σε, που ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική στρατηγική για την ισότητα των γυναικών και των αντρών που όπου θα λαμβάνει σοβαρά το υπόψη το ζήτημα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αναλαμβάνει ευθύνη. Αυτό σημαίνει επικύρωση και εφαρμογή τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη από όλου. Θα πρέπει η στρατηγική αυτή να περιλαμβάνει και την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, σεξουαλική εκμετάλλευση, προστασία και υποστήριξη των θυμάτων, ε, δίωξη των δραστών, και τα ευρύτερα δομικά ζητήματα να αντιμετωπιστούν, τα οποία προκαλούν αυτή τη βία. Θέλουμε να συνεργαστούμε λοιπόν με την Επιτροπή αυτή για την επικύρωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη ε, και για τι ευρύτερε στρατηγικέ, τι οποίε έγινε αναφορά. Χαίρομαι που είναι εδώ και οι δύο εισηγητέ. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σα για το θέμα αυτό. Ήρθε η ώρα. Υπάρχει πίεση, υπάρχει αυτή η ευκαιρία, υπάρχει πίεση από τι γυναίκε, από τα κορίτσια. Έχουμε δημιουργήσει την κατάλληλη πολιτική πίεση. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά και με αυτά θα δώσω το λόγο στην κυρία Τισέβα, Γενοβέβα Τισέβα, που είναι μέλος της Επιτροπής για την Εξάλληψη της Βίας των Γυναικών και θα μας μιλήσει της Επιτροπής για την εξέλιξη της βίας των γυναικών και θα μας μιλήσει για το τι διαδικασίες έχουν προβλεφθεί από την Επιτροπή αυτή για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, συνάδελφοι από τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και συνάδελφοι από διάφορες φορεί και την Κένια. Ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών και τη Ισότητα των Φίλων που με προσκάλεσε εδώ και μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω την δουλειά τη Επιτροπή μα για τη βία των ε, γυναικών τη χρονιά της, ε, την εξάλληψη των διακρίσεων στην 40η χρονιά επέτειο και επέτειο της λειτουργίας της. Εδώ μας ενδιαφέρει να φτάσουμε σε επέδο ισότητας και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών δίνοντάς τους τη δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτησίας, χειραφέτησης και να είναι ίσα μέρη, ε, οπότε όλα τα συμβαλόμενα μέρη και τα μέλη της Επιτροπής μας πρέπει να υιοθετήσουν ανάλογα μέτρα. Η ε, εφαρμογή της ε, σύμβασης της Επιτροπής μας που έχει οτιθεί από 113 χώρες μεταξύ των οποίων και κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο οδηγός μας. Οι βασικές ε, αρχές για την λειτουργία της σύμβασης είναι οι κατευθύνες γραμμές των κρατών μελών, οι εκθέσει που υποβάλλουν και η συνεργασία μας με τις κυβερνήσεις για το πώς λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Η διαδικασία follow-up ε, της παρακολούθησης είναι πολύ σημαντική για τη μέτρηση των φαινομένων βίας κατά των γυναικών να σας πω ότι πολύ συχνά οι εκθέσεις που φτάνουν στην Επιτροπή μας και όλη η διαδικασία συζήτηση των εκθέσεων αυτών στην εβδομάδα που συνεδριάζουμε είναι πολύ σημαντικά για να αναλυθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τη βία κατά των γυναικών. Στην πρόσφατη σύνοδο τη Επιτροπή μα ήταν σαφέ ότι η υλοποίηση των συστάσεων για τη βία κατά των γυναικών είναι θέμα προτεραιότητα για την παρακολούθηση από την Επιτροπή μα καθώς 36% των υποθέσεων και 5% των θεμάτων παρακολούθησης έχουν να κάνουν με την εξάλληψη ε, στερεοτύπων που αφορούν τα φύλλα και αρνητικών πρακτικών. Η ερμηνεία των διατάξεων της σύμβασης είναι σημαντικά για να συμπληρώσουν το διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίω τι βασικέ υποχρεώσει βάσει τη σύμβαση, καθώ και τη γενική, σύσταση 33, την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη από το 2013 και την σύσταση 35. 2017 για την έμφυλη βία κατά των γυναικών που ανταποκρίνεται και στη, σύμβαση, στη σύσταση 19. Οι νομικές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί βάσει και του πρωτοκόλου το οποίο ισχύει από το Δεκέμβριο του 2000 και έχει υιοθετηθεί από 113 χώρες ως τώρα είναι κάτι που θα πρέπει να προχωρήσει ταυτόχρονα με το μηχανισμό παρακολούθηση για να πάψει η, βία, η έμφυλη βία κατά των γυναικών και να περάσει αυτό και στο ε, εθνικό δίκαιο διεθνώ. Βασιζόμαστε σε δύο διαδικασίε. Ποινική διαδικασία που επιτρέπει οι ανακοινώσει τη Επιτροπή μα να ληφθούν υπόψη από συγκεκριμένα πρόσωπα ή ομάδα προσώπων σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων όπω καλύπτονται από τη Σύμβαση. Και μια άλλη διαδικασία που επιτρέπει η δική μα Επιτροπή να κινήσει διαδικασία για την ε, ε, διερεύνηση υπόθεση σε περίπτωση που προκύψει ε, περιστατικό κρούσμα παραβίαση γυναικών δικαιωμάτων. Εφόσον κρυφτεί το παραδεκτό ή όχι του αιτήματο, κοιτάζουμε κατά πόσο ένα κράτο μέλο έχει ε, σεβαστεί τι υποχρεώσει του βάσει τη σύμβαση. Και έτσι, αναλόγω, η Επιτροπή μα εκδίδει τι απόψει τη, αποστέλλοντας συστάσεις προς το για να αλλάξει την όλη κατάσταση με ένδικα μέσα που θα καλύπτουν τα δικαιώματα των ατόμων, των θυμάτων μεμονωμένα δηλαδή με την ανάλογη αποζημίωση και αποκατάσταση της ζημιάς, κάτι που ζητά συχνά η Επιτροπή μας, όπως και δομικές ή συστημικές αλλαγές που σκοπό έχουν να προλάβουν την ε, ε, εμφάνιση τέτοιων, την εκδήλωση τέτοιων παραβιάσεων και στο μέλλον. Εδώ λοιπόν θα πρέπει τα ατομικά δικαιώματα να προστατεύονται και τα δικαιώματα των γυναικών, η περίπτωση έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, η σεξουαλική βία, ο βιασμός, ε, η παραβίαση των δικαιωμάτων σεξουαλική και αναπαραγωγική υγείας, όλα αυτά να αντιμετωπίζονται επαρκώ. Έχουμε δει σε πολλά κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν στην νομοθεσία τους κενά που δεν επιτρέπουν να καλυφθούν αυτά τα δικαιώματα αρκετά. Θα ξέρετε την υπόθεση της Αυστρίας του 2005 όπου το, ο σύζυγος του θύματος πολλές φορές την είχε ξυλοκοπήσει και της είχε επιτεθεί με απειλές ε, κατά της ζωής της, κάτι που γνώριζαν η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές και είχε υποβληθεί και μήνυση, όμως ο εισαγγελέας την απέρριψε. Αυτό ε, το επιβεβαίωσαν και τα παιδιά τη. Είχε καλέσει την αστυνομία, είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία λίγε ώρε πριν δολοφονηθεί και τελικά δεν έγινε τίποτα. Η Επιτροπή μα λοιπόν, όταν παρακολούθησε την υπόθεση, ξέρει ότι την αγωγή την υπέβαλαν ε, τα παιδιά, οι στενοί συγγενεί τη ε, και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που οδήγησε στο να, αναλάβει η Αυστρία νομικές διαδικασίες για το θέμα αυτό, καθώς και νομική, δικαστική και οικονομική αρρωγή για όλα τα θύματα. Είχαμε κάποιες υποθέσεις από την Βουλγαρία, τον ε, υπόθεση VK ε, κατά Βουλγαρίας όπου δεν εκδόθηκε απόφαση ή εντολή προστασίας ασφαλιστικών μέτρων υπέρ του θύματος, θύμα από το οποίο είχε υπάρξει επανειλημμένα θύμα του συζύγου της, διότι τα γεγονότα της ε, βίας είχαν λάβει χώρα το μήνα προτού υποβληθεί η αγωγή. Η άρνηση του δικαστηρίου βασιζόταν σε στερεότυπα των φίλων, βάσει των οποίων ε, λειτουργήσε, και αυτό είναι κατά των ίδιων των ε, αρχών που διέπουν τη σύμβαση. Λοιπόν, η Επιτροπή μας θεώρησε ότι το δικαστήριο δεν πέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τα δικαιώματα των γυναικών βάσει των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει και με τη σύμβαση και αυτό θα πρέπει να, προλάβει, να αναλάβει μέτρα με επαρκή αποζημίωση για το θύμα βάσει και της ε, απόφασης του Συμβουλίου των Υπουργών και με αποζημίωση για άλλε δύο περιπτώσει παραβιάσεων δικαιωμάτων των γυναικών βάσει του σχετικού μα πρωτοκόλλου. Εδώ λοιπόν, ε, γι' αυτό το 2005 συγκεκριμένα, προβλέψαμε νομικό μηχανισμό για την οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση υποβολή ατομικών αγωγών. Τα γενικά μέτρα που σύστησε η Επιτροπή μα είναι πολύ σημαντικά και ήταν πολύ σημαντικά για τη συγκεκριμένη απόφαση αυτή ώστε να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης και να είμαστε βέβαιοι ότι ε, τα, του θύματος που μπορεί να υποβάλει η αγωγή θα εφαρμοστούν επιτέλους πράγμα που δεν είχε γίνει. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το παράδειγμα αυτό τη Βουλγαρίας είναι περίπτωση follow-up, παρακολούθηση του πώ εφαρμόστηκαν τα μέτρα, διότι η Επιτροπή ε, παρακολουθεί το πώς εφαρμόζονται τα μέτρα, τι μοτίβα εφαρμογής των μέτρων δημιουργούνται και τι continuum σε περίπτωση που το κάτω μέλος δεν έχει καλύψει όλα τα νομοθετικά κενά. Θα χρειαστούν λοιπόν εκεί τροπολογίες για να προστατευτούν οι γυναίκες σε περίπτωση οικονομική βία. Το 2014 η Βουλγαρία προσέφερε επιπλέον μέτρα ω πρόταση για την προστασία των σεξουαλικών δικαιωμάτων των γυναικών και το ίδιο και για ε, μία περίπτωση μίας ε, πολίτου από την Γκάμπια η οποία κατοικούσε εκεί. Εδώ λοιπόν σε περίπτωση τέτοιων ε, υποθέσεων, ακραίων υποθέσεων οικογενειακής βίας ή δολοφονίας των γενικών των παιδιών από τα παιδιά, ε, βάσει και τη ανακοίνωση 20 το 2011, ε, είχαμε μια ανάλογη περίπτωση και από τον Ανώτατο Δικαστήριο τη Ισπανία. Ήταν μια απόφαση πραγματικά καινοτόμα, πρωτοποριακή, γιατί το Ισπανικό δικαστικό σύστημα ε, κατα... κατέγραψε το δικαίωμα αυτών των γυναικών ω θεμελιώδε δικαίωμα βάσει και τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η κυρία Καρένιο είχε αφήσει το τριετές της παιδί, τον εγκατέλειψε αφού απείλησε τη ζωή τη και το ισπανικό δικαστικό σύστημα ήθελε να απαγορεύσει στην κόρη και να την ε, προστατεύσει από το να έχει δικαίωμα σε από τον βίο πατέρα ε, και αφού έγινε και, δικαστική, και έγινε ακρόαση στο δικαστήριο, ακρόαση της μητέρας, ήταν σαφές ότι θα έχανε την επαφή με την κόρη της ε, και αφού λήφθη η δικαστική απόφαση την επόμενη μέρα αυτοκτόνησε. Η δικαστική απόφαση συνεχίστηκε και κατόπιν αυτού αναγνωρίστηκε η ανικανότητα του κράτους να την προστατεύσει και να αναλάβει μέτρα ώστε να βεβαιωθεί ότι τα προηγούμενα γεγονότα ε, για την, ε, από την, της βία ε, έπρεπε να συμπεριληφθούν και να συνυπολογιστούν στο πώς θα κρυθούν τα δικαιώματα επίσκεψη του παιδιού. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε έκδοση σύσταση και την αλλαγή του ισπανικού νομικού συστήματος. Η, σύσταση λοιπόν της Επιτροπής μας ήταν υποχρεωτικού χαρακτήρα και το αναγνώρισε τελικά αυτό το ισπανικό δικαστικό σύστημα με ένα πολύ σημαντικό ε, πρόστιμο ε, αποζημίωση για την υπόθεση αυτή. Αυτά είναι απλώς μερικά παραδείγματα που δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν μέτρα κάποιες φορές και αναγνωρίζουν τα, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς ή διμερείς συνθήκες. Απλώς να πω ότι η Επιτροπή μας τονίζει τη σημασία του να ε, προσφέρουμε πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα και στη δικαιοσύνη για όλες τις γυναίκες ασχέτως εθνικότητας. Επίσης είναι σημαντικός ο ρόλος και η εξειδίκευση των δικηγόρων και των ε, δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και από διαφορετικά δίκτυα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και σε αυτό το πνεύμα οι συνάδελφοί μου από τη βουλγαρική υπηρεσία και τη δική μου ε, και επειδή είμαστε μέλη της Ανεξάρτητης Κοινωνίας των Πολιτών ξεκινήσαμε πριν από 15 χρόνια ένα πρόγραμμα, ε, ένα Ινστιτούτο εκπαίδευση σε συνάντηση, σε συνεργασία και με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Δικηγόρων ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες περιπτώσεις για το πρωτόκολλο και για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να συνειδητοποιήσουν επιτέλους τα κάτι μέλη ποιες οι υποχρεώσεις τους. Τελευταίο και εξίσου σημαντικό, η Επιτροπή ε, φροντίζει να επισημαίνει σχετικές υποθέσεις ε, όπου υπάρχουν κενά στην νομοθεσία των κρατών μελών για να προχωρήσουν σε κύρωση τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε συνεργασία και με την πλατφόρμα για την ανεξάρτητη παρακολούθηση της γενικής βίας και των δικαιωμάτων των γυναικών και τον ειδικό εισηγητή τον, του ΙΕ για τα θέματα αυτά, την κυρία Σιμόνοβιτς. Κοιτάζουμε λοιπόν το πώς η, η Επιτροπή μας ε, μπορεί να έχει ε, μια αρμονική συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τόσα προβλέπουν το Κοινοβούλιο και άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί για την προστασία των ε, γυναικείων δικαιωμάτων προκειμένου να αποφύγουμε και άλλες περιπτώσεις θανάτων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας μπορούμε πραγματικά κάτι να κάνουμε και να γίνει μια διαφορά. Έχουμε πολλά εργαλεία. Ο λόγος τώρα σε εσά. Πρώτα ο λόγος στην εισηγήτρια, την κυρία Κοκολάρη. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Άλβα Κοκολάρη και είμαι ε, νέο μέλος ε, του Κοινοβουλίου από τη Σουηδία μια από τις χώρες που θεωρείται μια από τις ε, πρωταθλήτρες της ισότητας των γυναικών στον κόσμο, αλλά και εμείς έχουμε προβλήματα όπως τα ξέρετε. Το ξέρετε εσείς, ε, κυρία μου, και εδώ είμαι συγγήτρια για τα θέματα της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Είμαι πραγματικά ταγμένη στο σκοπό αυτό, προκειμένου να γίνει πρόοδο στο θέμα και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας θα καταφέρουμε να έχουμε ευρωπαϊκό νομοθέτημα, δηλαδή ευρωπαϊκή προσχώρηση στη σύμβαση. Πιστεύω ότι τελικά όλα τα κράτη-μέλη θα την κυρώσουν και νομίζω ότι αυτό θα είναι μια πραγματική επιτυχία για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη. Αλλά και ένα σαφέ μήνυμα για όλο τον κόσμο ότι η Ευρώπη δεν θα ανεχτεί άλλο τη βία κατά των γυναικών. Πρέπει να κάνουμε τα εξή δύο. Πρώτα απ' όλα να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση θα το πράξουν αυτό ως το δυνατόν συντομότερα και ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και από την πλευρά των άλλων κατομελών να μάθουν ότι όσοι δεν την έχουν κυρώσει ότι η βία και τα ε, σοβαρά εγκλήματα δεν είναι αποδεκτά στην Ένωσή μας και πρέπει να εξαλειφθούν ε, και στην περίπτωση των γυναικών που είναι τα θύματα. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας αρέσει να λέμε ότι τα προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι η θεμέλιά μας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αξίες του ανθρωπισμού, όμως δεν σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ένωσης πολλέ φορέ. Γι' αυτό λοιπόν δική μα ευθύνη είναι εμεί ω νέοι βουλευτέ και ελπίζουμε το ίδιο θα κάνει και η Νέα Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουμε περισσότερο για να προστατεύουμε όντω τι θεμελιώδει αξίε και τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτά πραγματικά θα έχουν ένα υψηλό επίπεδο σεβασμού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπω έχω πει όλοι, θέλουμε να υπάρξει κύρωση. Κύρωση σε ευρωπαϊκή. Επίση, τα θύματα τη εμπορία των σεξουαλικών εγκλημάτων θέλουμε και αυτά να προστατεύονται. Θέλουμε λοιπόν η έμφυλη βία να συμπεριληφθεί ω ένα ε, χώρο ποινικού δικαίου ε, και να καλύπτεται. Ε, θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε θετικό διάλογο, επικοδομητικό μεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερομένων και των διαφόρων πολιτικών ομάδων και θα πρέπει να ε, πιέσουμε και τα κατημέλη και το Συμβούλιο για να κάνουν κάτι. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει συζήτηση για την σύμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο και πραγματικά ανυπομονώ για τη διεξαγωγή της συζήτηση αυτής. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε να συζητιέται το θέμα αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο και είμαι και βεβαίω ότι η Ursula von der Leyen που έχει δεσμευθεί ότι θα αναλάβει δράση για τα θέματα αυτά θα την πιέσουμε και εκείνη. Και το νέο Ευρωκοινοβούλιο με πολλά νέα μέλη που είναι πρόθυμα να αγωνιστούν για μια καλύτερη Ευρώπη μια Ευρώπη όπου τα θεμελίδια δικαιώματα θα καλέπτονται. Ελπίζουμε ότι κάτι θα καταφέρουμε. Έχω δύο ερωτήσει προ τον Γκρέβιο, την οργάνωση Γκρέβιο. Ε, για παράδειγμα, στη χώρα μου τη Σουηδία, όπου η ισότητα των φύλων είναι πραγματικά ένα θέμα στο οποίο όλοι δείχνουν σεβασμό. Έχουμε ένα νέο φαινόμενο, την ψηφιακή βία. Βλέπουμε σεξουαλική παρενόχληση να παίρνει διαστάσει επιγραμμικά online το Γκράβιο, τι ε, μπορεί να κάνει για το φαινόμενο αυτό, τι προτείνετε εσεί για το τι μπορεί να γίνει στο ίντερνετ για την σεξουαλική παρενόχληση και τη βία κατά των γυναικών, φαινόμενα που παίρνουν διαστάσει και έχουν διεγκωθεί στο διαδίκτυο και πώ επίση μπορούμε να οργανώσουμε τη ε, συνεργασία μα με άλλα κρατημέλη και οργανισμού, ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσει για το περιεχόμενο τη σύμβαση. Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να πέσουν τα ταμπού σε συγκεκριμένα κρατημέλη. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σπούρεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ξέρετε είμαι μία από τις δύο συγγήτριες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό ε, της ε, προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση ε, της Κωνσταντινούπολης το οποίο είναι απαραίτητο να συμβεί. Ε, ένα ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συζήτηση της επόμενης εβδομάδας για να κάνει με τα δύο φύλλα. Ε, όλα τα κράτη-μέλη αποδέχονται ότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ε, τα δύο φύλλα σε ό,τι αφορά ε, την κατανομή των κονδυλίων αλλά δεν λαμβάνεται αυτό υπόψη σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών και την ενδοκοινωνιακή βία. Μίλησα με την πρόεδρο νωρίτερα γι' αυτό. Θα πρέπει πραγματικά να υπογραμμίσουμε ότι η Σύμβαση Κωνσταντινούπολη ε, έχει να κάνει με το να σώζουμε ζωές. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Ένα σχόλιο είναι από, το, από την πλευρά μου. Ευχαριστώ η κυρία Κάνκο που την κυρία Άντερσον. Thank you very much. I would like to repeat... Ευχαριστώ. Ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε η κυρία Μέικοκ. Είπε ότι δεν υπάρχει ειρήνη όταν η γυναίκα φοβάται για την ασφάλειά τη στο σπίτι τη και στο δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών και εδώ στο Βέλγιο, στη χώρα μου, αλλά και στη χώρα προέλευσή μου, τι λέει ο κόσμο, Ναι, σημειώνουμε πρόοδο, βελτιωνόμαστε. Μπορεί να φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά τη γυναίκα η οποία ε, ζει τη βία στο σπίτι τη, δεν προχωράμε από τη δική της οπτική γωνιά. Πρέπει να σκεφτούμε πάντα αυτούς οι οποίοι δεν βλέπουν αυτή την πρόοδο. Αυτό που με ανησυχεί, είμαι και η εισηγήτρια για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από την ομάδα ECR, είναι ότι συχνά επαναλαμβάνουμε αυτά που ακούμε για τα δικαιώματα των γυναικών. Έχω πάει σε τόσες ακροάσεις, ε, σε διασκέψεις, σε συζητήσεις και υπάρχει πολλή βία. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα. Τι θα κάνουμε στις επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Πώς θα δώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό, όχι απλώς να περιγράφουμε ξανά και ξανά τη κατάσταση. Äh, Frau Maria Neuchel. Ευχαριστούμε. Ε, και τώρα η κυρία Νόιχλ. Η κυρία Άντερσον μάλλον και μετά η κυρία Νόιχλ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα σημεία. Μιλήσατε για το stalking, την επίμονη παρενόχληση αρχίζουμε να έχουμε όλο και περισσότερους νόμους για αυτά. Εγώ είχα ζήσει εκείνο το διάστημα στις ΗΠΑ και ήταν πολύ ε, σημαντικό το ότι η αστυνομία που γνώριζε περιπτώσεις γυναικών που ήταν θύματα παρενόχλησης δεν είχε κάνει τίποτα και τελικά τις έβρισκαν ακραίες. Η σεξουαλική λοιπόν παρενόχληση είναι το επόμενο θέμα. Η παρενόχληση των γυναικών στον εργασιακό του χώρο. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα. ίσως από αβεβαιότητα το ποιος, τι και γιατί και πώς αυτά μπορούν να αξιολογηθούν. Τότε το πρόβλημα της, των ΗΠΑ ήταν το τι θα γίνει με την ε, πολιτική που εφαρμόζεται την ιδιαίτερη ενεκτικότητα που έδειχναν για τα διευθυντικά στελέχη και το κατά πόσον αυτοί που ασκούσαν τη σεξουαλική παρενόχληση είναι του πιο κοντινούς των γυναικών αυτών. Η ερώτησή μου λοιπόν αυτή είναι το κατά πόσον υπάρχει η πιθανότητα από τη μια οι πολιτικέ τη σεξουαλική παρένόχληση όντω να προβλεφθούν και να εφαρμοστούν και από την άλλη να κάνουμε κάτι έχοντας σε κάθε περίπτωση δυνατότητα καταγγελία και σε μια συζήτηση χωρί φραγμού με του συναδέλφου στον εργασιακό χώρο. και για το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Έχουν γίνει αξιοσημείωτα βήματα πρόοδου, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρούμε ότι υπάρχει και μια οπισθοδρόμηση πολλές φορές για την ενδοοικογενειακή βία στην ε, Γερμανία. Βλέπουμε να υπάρχει ένα apartheid ε, με βάση τα φύλλα. Ε, Φαίνεται δηλαδή ακόμη και στον δημόσιο χώρο να μην υπάρχει απόλυτη προστασία των γυναικών που μπορεί να έχουν ε, περιπτώσεις σεξουαλικής ε, βίας εναντίον τους και η αστυνομία να μην αναλαμβάνει δράση. Να ρωτήσω μήπως αυτό είναι μια νέα περίπτωση του victim blaming όπως το λέμε δηλαδή ότι αντιστρέφεται η θέση του θύματος και κατηγορούνται τελικά οι γυναίκες που υπήρξαν θύματα είναι κλασικό η περίπτωση. Ξέρουμε την πρόσφατη περίπτωση που προκύψε στο διαδίκτυο με 106 παιδιά που ήταν θέματα, θύματα ε, βιασμών και σεξουαλικής ε, κακοποίησης. Ε, μιλάμε για την περίπτωση γυναικών, νεαρών κοριτσιών μάλλον, που ήταν τέτοια θύματα σεξουαλικής βίας. Εδώ λοιπόν ε, υπάρχουν σοβαρά βήματα πρόοδου που πρέπει ακόμη να γίνουν. Εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι ώστε ιδεολογικά σε περιπτώσεις ε, και ισλαμικής διείσδυσης δεν καλλιεργούνται περαιτέρω στερεότυπα στην Ευρώπη. Και εάν έπρεπε να αποτιμήσετε αυτή την κατάσταση για τις μουσουλμάνες, ε, για τους πιστούς του Ισλάμ, τι θα μπορούσατε να προτείνετε, τι συστάσεις να υπάρξουν και προκειμένου να προστατευτεί και η ζωή τους. Τι νομικέ, νομικά μέτρα θα πρέπει να υπάρξει μια διάκριση βάσει των θρησκευτικών πεπιθήσεων και οι γυναίκες αυτές να αναγνωριστούν ως προς και τη σεξουαλική τους, ε, την ανάγκη για τη σεξουαλική τους προστασία και τη σωματική ακαιρεότητα. Ευχαριστούμε κυρία Νόχλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω αλλά έχω διαφορετικές ερωτήσεις από την ομιλητριά μας, ε, από την προηγούμενη ομιλητρία. Ξέρουμε ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει γίνει, έχει κυρωθεί από κάποια κάτι μέλη, αλλά κάθε ένα κάτω μέλος που έχουμε πετύχει να κυρώσει είναι μια επιτυχία και κάνουμε ένα τικ στον κατάλογο των κρατών που το έχουν πράξει αυτό τώρα για τη Γερμανία. Ήθελα να μου πείτε τις συγκεκριμένε απόψεις σας για το πώ γίνεται από τη μια, μια χώρα στην Γερμανία να έχει υπογράψει τη σύμβαση αυτή και να την έχει κυρώσει και από την άλλη ε, να παραμένουν υποχρεώσει στο χαρτί. Και μόνο. Διότι οι γυναίκες ε, ε, στη Γερμανία ουσιαστικά έχουν τη δυνατότητα να ε, στην ουσία οι γυναίκες στη Γερμανία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, πρώτη και δεύτερη. Τι πρέπει να γίνει με τις γυναίκες που προέρχονται από άλλη χώρα είναι δυνατόν ε, γυναίκες διαφορετικής εθνικότητας στην ίδια χώρα να τη χάνουν διαφορετικής μεταχείρισης και να έχουν διαφορετικά δικαιώματα. Οι Ρουμάνες, ας πούμε, οι οποίες εκπορνεύονται στην ε, Γερμανία, δουλεύουν σε αυτόν τον ε, τομέα, στη Γερμανία δεν έχουν άλλα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι μία ε, διακριτική μεταχείριση και το θέμα δεν είναι απλώς να βάζουμε το τίξτο κουτί της κύρωσης, αλλά να ξέρουμε ότι όλα εφαρμόζονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Η τελευταία συνάδελφο τώρα, κυρία Φιτζέραλτ, και μετά η ομιλήτριά μα για να απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Με τρομοκρατούν τα δεδομένα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αντίσταση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό που μου έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση από τότε που έχω γίνει μέλος εδώ και ακούω τις γενικότερες συζητήσεις είναι όλες αυτές οι προβολές ό,τι αφορά τη σύμβαση. Βεβαίως έχει να κάνει με τη βία ενάντια στις γυναίκες και παρόλα αυτά έχουμε αυτές τις ιδεολογικές προβολές και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτησή μας. Πρέπει να έχουμε μια υψηλού επίπεδου στρατηγική, μια πολιτική συζήτηση για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε το ζήτημα αυτή, αυτό. Γνωρίζω ότι αυτό κάνετε όλη την ώρα, δεν, λέω ότι είναι απλό, αλλά πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Σε αρκετές χώρες υπάρχουν καινούριε νομοθεσίε, υπάρχουν πρωτοβουλίες κτλ. κτλ. Είναι όμως ένα τόσο τρομερό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Μόλις έρχομαι από τον Αιρόμπι, από μια συνεδρίαση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του πληθυσμού και όλα αυτά τα οποία πρέπει να υπομείνουν οι γυναίκες, έτσι όπως τα άκουσα εκεί, είναι πραγματικά τρομερό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε μια υψηλού επίπεδου στρατηγική. Μια συνάδελφος ήδη το είπε, πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή της λύσης και όχι να περιγράφουμε το πρόβλημα. Και αυτό πιστεύω κι εγώ. Υπάρχουν λύσεις σε ό,τι αφορά τη βία στον κυβερνοχώρο, το τράφικινγκ κτλ. Η εφαρμογή όμως, το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια αυτά, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Υπάρχουν ευκαιρίες αυτή τη στιγμή. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ το να περιγράψουμε την υψηλή επίπεδο δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε. Και θα ήθελα επίσης να προτείνω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να συζητήσουμε με άτομα που δεν εκτίθενται σε τέτοιου τύπου συζητήσεις συνεχώς. Το, το να μιλάμε, υπάρχει τάση να συζητάμε τα θέματα ισότητας με τους ίδιους και τους ίδιους. Είναι ένα πρόβλημα που έχουν και αυτές οι επιτροπές εδώ πέρα. Πρέπει όμως να μιλήσουμε στα άτομα που αντιστέκονται, στα άτομα που αντιστρατεύονται τις αλλαγές είναι ένα τεράστιο έργο που θα πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή αυτή ε, το χρόνο που έρχεται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ένα στρατηγικό έτος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Τα εμπόδια όμως, ιδίως ό,τι αφορά την ιδεολογία, είναι πολύ ισχυρά. Και ανησυχώ ότι μπορεί να μην είναι εύκολο να τα ξεπεράσουμε. Με ενδιαφέρει όμως να ακούσω ποια είναι η άποψή σας, το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ε, κυρία το λέει και μετά κλείνω κατά I will try to be the, the positive uh, speaker. It's... Uh, θα προσπαθήσω να μιλήσω κάπως ε, θετικά. Είναι ήδη καλό ότι έχει υπογραφεί και επικοινωθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από τόσες χώρες. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να πείσουμε ε, τις χώρες που ακόμα αντιστέκονται, ιδίως τις ευρωπαϊκές χώρες διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ε, στην πρώτη γραμμή σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως ε, είχαμε ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο στην Γαλλία για το θέμα αυτό. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη αναγνώρισε ε, ότι δεν ξέρει πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα. ο δρόμο ο, ο νόμος μάλλον μπορεί να αλλάξει, αλλά το θέμα είναι πώς γίνονται περιγραφέ στη συνέχεια από τι αστυνομικέ αρχές πώς εξετάζονται στο δικαστήριο. Πρέπει να αλλάξει συνολικά η θεώρησή μας το πώ προσεγγίζουμε τα ζητήματα αυτά για να είναι αποτελεσματικά, αυτέ οι αλλαγέ. Μου έκανε πραγματικά εντύπωση ιδιαίτερα το θέμα των παιδιών διότι όταν μια γυναίκα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, έχει υποστεί βία, ε, επειδή κρατάει το παιδί, μένουν μαζί και είναι σε κίνδυνο μαζί. Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να προστατεύει την οικογένεια από τη βία μετά την πρώτη πρώτο κρούσμα χωρίς αυτή την ιδέα ότι πρέπει όλοι να ζουν μαζί ε, δηλαδή και ο δράστης ε, ο οποίος μπορεί να επανέλθει είναι ο λόγος της γυναίκας απέναντι στο λόγο του άντρα, λέει η αστυνομία. Τι κατάρτιση, τι εκπαίδευση έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ αυτό που θα ήθελα θα ήταν όλες οι καλές πρακτικές που υπάρχουν στην κάθε χώρα να τις μοιραστούμε για να διευκολύνουμε την εφαρμογή της Σύμβασης της Ισταμπούλ για όλα τα κρατημέρια για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών στην Ευρώπη ε, και δυνατόν και στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ και τους τρεις σας για τις καταπληκτικές παρουσιάσεις, λέει η Τζάκι Τζόουνς. Ευχαριστούμε πολύ ε, και την προσπάθειά σας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς. Εγώ είμαι νομικός και με ενδιαφέρει η νομοθεσία. Και αυτά που είπατε για τις νομοθεσίες και τις πολιτικές αν τα κατάλαβα καλά, ε, αυτό που αναφέρονται στην έκθεση της Γκρέβιους ε, και στις συστάσεις ε, ε, αναφέρεστε στις παρεμβάσεις τρίτων. Ε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή Γυναικών για να βοηθήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό χρειάζεται χρήση χρηματοδότησης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε κατά πόσο, δεν, έχω, δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό, ε, γίνεται μια συζήτηση για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να δοθούν κάποια κονδύλια για παρεμβασει ε, τρίτων ή για ε, συλλογικές ε, προσφυγές ε, και αν επιθυμείτε κάτι τέτοιο βέβαια εσει Σε ό,τι αφορά το πω συνδέεται η νομοθεσία με τις πολιτικές σε σχέση με αυτό που ρώτησε και η Μαρία ε, για τι γυναίκε μετανάστριες και τι γυναίκε που, έχουν ένα, που ζουν σε ανασφαλέ καθεστώ, υπάρχει ο χάρτη, ε, η Χάρτα Μελιών Δικαιωμάτων που εφαρμόζεται σε όλου όσου βρίσκονται εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. έτσι. δεν εξαρτάται από την ηθαγένεια η χάρτα αυτή εφαρμόζεται σε αυτού. αυτό λοιπόν συνδέεται με μια χρηματοδότηση που θα μπορέσει να βοηθήσει με με την εφαρμογή στα πλαίσια της, ε, του χάρτη των δικαιωμάτων μαζί με τη σύμβαση της Ισταμπούλ και βεβαίω υπάρχει και το Συμβούλιο της Ευρώπη με 47 του μέλη. Ε, ευχαριστώ για όλες αυτές ε, τις ερωτήσεις και για όλα αυτά τα πολύ σωστά ερεθίσματα που θέσατε. Τώρα θα δώσω το λόγο στις προστεκλημένες μας. Κυρία Νάουντι, αν θέλετε ξεκινήστε. Έχετε πολλά ερωτήματα. Πρέπει να έρχομαι ίσως πιο συχνά, ούτως ώστε σιγά σιγά να απαντήσω στα ερωτήματά σας. to, okay, violence. Το, το ζήτημα της βίας στον κυβερνοχώρο, πρώτα απ' όλα, και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα που διαρκώς διωγγώνεται. Εξής όμως διωγγώνεται και η γνώση που έχουμε πάνω στο ζήτημα αυτό. Αν κάποιος με παρενοχλεί στο δρόμο, αν κάποιο με παρακολουθεί στο δρόμο ή αν κάποιο με παρακολουθεί στο διαδίκτυο, θα πρέπει να υπάρχει ένα νόμο που να με καλύπτει. Αν κάποιο με παρενοχλεί σεξουαλικά στο χώρο εργασία μα, ή αν κάποιο με παρενοχλεί ε, σεξουαλικά στο διαδίκτυο, θα πρέπει να υπάρχει ένα νόμο που με καλύπτει. Επομένω, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα, το πρώτο σημείο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Παρ' όλα αυτά όμω, όπω είπα και προηγουμένω, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη προσοχή σε ό,τι αφορά στη βία στο διαδίκτυο, σε ό,τι αφορά την έντονη παρακολούθηση και κάπως αλλιώς αποκαλείται, αλλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Και η ομάδα μας το Γκρέβιο θα συμμετάσχει σε μια συνάντηση που θα γίνει το Δεκέμβριο πάνω στο ζήτημα αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να έχουμε μια κοινή θέση ούτω ώστε να παρακολουθήσουμε τις διαφορετικές χώρες με τις οποίες το έχουμε συζητήσει και να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τι δρόμο θα ακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την παραπληροφόρηση, τις παρερμηνίες και το τι μπορούμε να κάνουμε, το είπα και προηγουμένως, θα το ξαναπώ. Βγείτε έξω, ιδίω αυτές τις χώρες όπου ήδη έχουν γίνει κάποιες αλλαγές εξαιτίας της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αλλαγές προς το καλύτερο. Οι, οι χώρες αυτές που έχουν αξιολογηθεί και έχουν δει τις ε, θετικές επιπτώσεις της αξιολόγησης. Βγείτε έξω και πείτε το, επικοινωνήστε το. Γιατί αυτοί που διαδίδουν ε, λάθος πληροφορίες ουρλιάζουν. Και πρέπει να φωνάξουμε και εμείς εξίσου. Πρέπει και εμείς να ουρλιάξουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας, ούτως ώστε να ακουστούν και τα θετικά πράγματα. Όχι μόνο εδώ μεταξύ μας και εκεί έξω. Πρέπει λοιπόν να βγούμε στο, στο δρόμο, να επικοινωνήσουμε ε, με όλο τον κόσμο. Δυνατά, ενωμένοι, πρέπει να κάνουμε θόρυβο. Υπόθηκε επίσης κάτι σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε προς τα μπρος, γιατί κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι πάμε προς τα μπρο, αλλά υπάρχουν γυναίκες που βρίσκονται ακόμη σε πολύ δύσκολη κατάσταση και υπάρχει αυτή η έκφραση «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω». Αυτό κάνουμε, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Πρέπει να παλέψουμε για όλες τις γυναίκες. Όχι μόνο για να έχουμε μια καλύτερη θέση εργασίας, αλλά και για αυτές τις γυναίκες που βρίσκονται σε τελείως διαφορετικέ καταστάσεις. Θέλω να σας πω απλά. Οι πισίνες, ξέρετε, εγώ έρχομαι από μια εποχή που υπήρχαν πισίνες. Υπάρχουν πισίνες που είναι μικρές. Αλλά α, μπορούν να δημιουργήσουν τεχνητά κύματα, ούτω ώστε να μπορεί κανείς να κολυμπήσει κόντρα στο ρεύμα, χωρίς να βρίσκεται σε μια τεράστια πισίνα. Και κάποιο μου είπε πρόσφατα, όταν έλεγα, κοίτα, γέρασα και παλεύω ενάντια στη βία ενάντια των γυναικών και καμιά φορά αισθάνομαι δεν έχω κάνει ούτε μισό βήμα προς τα μπρος. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, σκέφτομαι ότι αν δεν παλεύαμε όλα αυτά τα χρόνια θα μας είχε πάρει το ρεύμα προς τα πίσω και ακριβώς επειδή τόσα χρόνια παλεύουμε μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο προς τα μπρος και αν δεν παλεύαμε θα μα έπαιρνε το ρεύμα, γι' αυτό δεν τα παρατάμε, γι' αυτό συνεχίζουμε να παλεύουμε. Πώς να αξιολογήσουμε τη σεξουαλική ε, παρενόχληση στο χώρο εργασίας, να το ξεχωρίσουμε από ένα «θες να πάμε για καφέ». Λοιπόν, εγώ ε, επιτρέψτε μου να σηκωθώ. Και εγώ δουλεύω σε ένα πανεπιστήμιο, είμαι ακαδημαϊκός. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σηκωθώ. Λέω στους φοιτητέ μου. Είναι ένα πράγμα να έρθει κάποιο και να σου πει «Καλημέρα» και κάτι άλλο να πλησιάσει, να σκύψει προς το μέρος σου και να σου πει «Καλημέρα». Το δεύτερο είναι σαφέστατα σεξουαλική παρενόχληση. Το πρώτο, όχι. Επιπλέον, αν το, απλά και μόνο το γεγονό ότι λέω σε κάποιον καλημέρα σε μια γυναίκα, τότε η γυναίκα αυτή έχει το δικαίωμα να μου πει μου κάνει τη χάρη, σε παρακαλώ, με ενοχλεί όταν οι άνθρωποι με πλησιάζουν. Και εκεί θα πρέπει να τελειώνει η υπόθεση αν όμως κάποιος αντιδράσει και πει με αυτές οι γυναίκες δεν μπορούσε να τους πείσετε μια καλημέρα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι σαφές, με άλλα λόγια. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο πότε υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ως γυναίκες μας έχουν πει, έχουμε αποδεχτεί, έχουμε απορροφήσει την πραγματικότητα ότι μπορεί κάποιος να μας παρενοχλήσει. Πολλοί γυναίκες λοιπόν σηκώνονται και λένε αρκεί, φτάνει, δεν θέλω. Γιατί μεγαλώσαμε με τον τρόπο του, από αυτό το να περιμένουμε σεξισμό κάθε μέρα, παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Γι' αυτό το λόγο το αποδεχόμαστε. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να μάθουμε από την αρχή, μάλλον να ξεμάθουμε όλα αυτά που μας έχουν πει και να πούμε στον εαυτό μας αξίζω, έχω αξία και δεν θα επιτρέψω κανέναν να μου συμπεριφέρεται με έναν αρνητικό τρόπο. Θεωρώ ότι αυτό είναι μέρος της απάντησής σας. Υπήρχε και ένα ερώτημα για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, ένα σχόλιο. Και πάλι, υπάρχει κι άλλο ένα ρητό που λέει ότι όταν δείχνεις τον, ε, τον γείτονά σου με το δάχτυλο, τότε κάποιος θα σε πυροβολήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο. Έχω βρεθεί σε άλλες χώρες και μου έχουν πει ότι δεν έχουμε την παράδοση του να δέρνουμε τις γυναίκες μας. Και εγώ λέω, ήμαρτον. ποιο έχει την παράδοση να δέρνει γυναίκες. Υπάρχουν όμως χώρες που οι άντρες χτυπάνε τις γυναίκες. Με συγχωρείτε, αλλά παθιάζομαι. Ε. Γιατί είναι άδικο. Γιατί δεν θα πρέπει να το αποδεχτούμε. Είναι ανάγκη να πούμε φτάνει, αρκεί, όχι. Ε, άτομα που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι μια χώρας δεν καλύπτονται. Καλύπτονται σύμφωνα με τη συνθήκη της, ε, τη σύμβαση με συγχωρείτε, της ε, Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγέ που μπορούν να κάνουν οι χώρε όταν επικυρώνουν την σύμβαση. Αυτό όμως που λέμε ότι η άδεια παραμονής κάποιου που εξαρτάται από το σύντροφό του και είναι, σύντροφό και είναι θύμα βία από το σύντροφό τότε μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη κάτοικος από μόνη της αν εγκαταλείψει το σύντροφο. Εκεί είναι το πρόβλημα, η επιφύλαξη που έχουν ε, θέσει κάποια κράτη. Όμως επί της ουσίας καλύπτονται από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Κάποια κράτη έχουν αυτή την επιφύλαξη ότι οι γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν από μόνος τους άδεια παραμονής και γι' αυτό το λόγο εξαρτώνται από το σύντροφο. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα για τα παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά θα αφήσω και κάποιον άλλο να μιλήσει γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να δώσω τώρα το λόγο. Είναι τόσο συναρπαστικό να σας ακούμε και είναι τόσο εμψυχωτικά αυτά που μας λέτε που έχουμε καθυστερήσει στην ακρόασή μας αλλά πρέπει να ακούσουμε και τι προκεκλημένε μα με τι απαντήσει του, όσο δυνατόν πιο σύντομο, παρακαλώ. Αυτό δείχνει πόσο ενδιαφέρον υπάρχει και δείχνει και πο... γιατί πρέπει να το κάνουμε και πιο συχνά. Ε, σέβομαι βεβαίω ότι υπάρχει και, και άλλο πάνελ, οπότε θα είμαι σύντομη. Ε, είμαστε εδώ εμεί ω Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών. Έχουμε μέλη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε και εδώ στι Βρυξέλλε. Αν οποιοδήποτε θέλει να συζητήσει μαζί μα για το έργο μας, για την ανάλυση μας, τις ιδέες μας για το μέλλον, ξέρετε που να μας βρείτε. Θέλω μόνο να πω τρία πράγματα, πολύ σύντομα. Πρώτον, κάτι που είναι ζωτική σημασία για αυτή την Επιτροπή. Ένα από τα πιο δύσκολα ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολη ε, Κωνσταντινούπολης είναι ότι εξαρτάται πού βρίσκεται μια γυναίκα και τι πρόσβαση έχει στη δικαιοσύνη, εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία, εξαρτάται από τι αστυνομικέ αρχέ, εξαρτάται από τη χώρα, εξαρτάται από πολλέ και διάφορε διακρίσει τι οποίες μπορεί να αντιμετωπίζει. Και αυτή η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επανειλημμένως έχει πει ότι αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να μπορεί μια γυναίκα να κολλήσει όπου και να πάει, να έχει την ίδια πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την ίδια υποστήριξη, τα ίδια δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει αυτό και γι' αυτό χρειάζεται μια συνολική, σφαιρική ευρωπαϊκή δράση. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να λάβουμε δράση. Να μην μιλάμε μόνο για το πρόβλημα. Αλλά είναι αλήθεια ότι και πολλοί δεν αντιλαμβάνονται το εύρος του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Πόσο δηλαδή, ε, πόσο μεγάλο πεδίο καλύπτει. Ε, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό για να βρούμε τις λύσεις. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη γραμματεία του Συμβουλίου εδώ στις Βρυξέλλες, με εσά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα με τους εισηγητές ε, και τα μέλη της Επιτροπής αυτής, ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και με άλλες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, δημιουργούμε μια συμμαχία και με τα συνδικάτα έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίζουμε να, βρούμε, να βρίσκουμε λύσεις και να πιέζουμε για την πλήρη επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Ε, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει άλλη μια συλλογή υπογραφών για να υπάρξει δημόσια υποστήριξη για αυτό το δημόσιο αίτημα σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει πίεση σε χώρες ε, όπου υπάρχει υποστήριξη αλλά δεν πιέζουμε αρκετά τις χώρες που μας κρατάνε πίσω. Η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες χώρες πρέπει να πιέσουν. Θα δώσουμε λοιπόν έμφαση σε αυτή τη μορφή πίεσης, ε, σε αυτή τη φάση. Ξέρουμε ότι αυτή η Επιτροπή θα μας υποστηρίξει. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας υποστηρίξει γενικότερα ε, για να σταματήσει, να βάλουμε τέρμα ε, στη βία κατά των γυναικών και να δημιουργηθεί ένα πλήρε νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την εξάλληψη τελικά τη βία κατά των γυναικών. Ένα πράγμα είναι η επικύρωση και εφαρμογή τη ε, σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα όμω έχει έρθει η ώρα να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οδηγία για τη βία κατά των γυναικών. Νομοθεσία, ενισχυμένη νομοθεσία για την καταπολέμηση τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και των κοριτσιών. Και αυτό πλέον έχει διαστάσει επιδημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι. Η Τζάκη αναφέρθηκε ε, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία, όμως ε, είναι και οι οργανώσεις των γυναικών, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που εργάζονται εκεί, στην πρώτη γραμμή, ε, για να βάλουν τέλος στη βία κατά των γυναικών. Επίση χρειαζόμαστε καλύτερα και περισσότερα δεδομένα. Θα αναφερθεί στη συνέχεια η ΆΙΝΤΑ, που έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια ε, ιδιαίτερα η δουλειά που γίνεται για τις γυναικοκτονίες και κάτι τελευταίο για την βία στο διαδίκτυο. Συνεργαζόμαστε με τα μέλη μας για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ε, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, κοινή κατανόησης. Όπως είπα, αυτό αποτελεί μέρος ε, της ευρύτερης, βίας κατά των γυναικών. Ε, επίσης, στις ευρωεκλογές συνεργαστήκαμε με τα πολιτικά κόμματα και με τους πολιτικούς θύνοντες, διότι ανησυχούμε ε, για το πώς ε, τελικά αυτή η βία στο διαδίκτυο ε, θέτει στο στόχαστρο γυναίκες της πολιτικής, γυναίκες υποψηφίους, γυναίκες που μιλάνε για τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι άλλος ένας τρόπος για να φημώσει κανείς τις γυναίκες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε μαζί σας και για αυτές τις πτυχές της βίας στο διαδίκτυο κατά των γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα της πολιτικής αλλά και γενικότερα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ε, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό κατά τη γνώμη μας. Χρησιμοποιείται επίσης όλο και περισσότερο ως τρόπος ε, οργάνωσης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών επιγραμμικά μέσω της πορνογραφίας, ε, του grooming, μέσω της εμπορίας ανθρώπων μέσω της πορνείας. Πρέπει λοιπόν μια ευρύτερη, να λάβει μια ευρύτερη πολιτική δράση για τα ζητήματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, τελευταία ομιλήτρια αυτού του πάνελ, η κυρία Τίσεβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα επαναλάβω αυτά που έναμε οι συνάδελφοι και θα ολοκληρώσω και με μία έκκληση. Περισσότεροι άντρε πρέπει να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα και θα πω και γιατί γιατί και για εκείνου είναι όφελο να καταπολεμηθεί αυτή η ιδεολογία. Πρώτα απ' όλα, στην ε, Επιτροπή μα βλέπουμε ότι όλα τα θέματα αυτά είναι εντελώ αλληλένδετα και είναι μια διαδικασία πολύ επώδυνη προκειμένου να πείσουμε και όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσουν τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Δεν θα πω πόσο καλά γνωρίζω την κατάσταση στο πετσί μου και τι έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα μου. Απλώ αυτό που είπαμε για την ε, ε, Επιτροπή μας και το τι γίνεται στις διαφορετικές χώρες. Πώς έχουμε δει να υπάρχει επιδείνωση και υποβάθμιση των δικαιωμάτων και όσων προβλέπει το άρθρο 5 για την υποβολή εκθέσεων για τα θέματα στερεοτύπων των φύλων και τις επιζήμιες πρακτικές. Τέτοιου είδους πρακτικές πραγματικά ε, ανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πραγματικά, αυτή η οπισθοχώρηση, αυτή η οπισθοδρόμηση μάλλον, είναι κάτι το επώδυνο και για την Επιτροπή μα. Και εκθέσει των κατομέλων για, για την έμφυλη βία, ακόμη και αν έχουν κάποια βήματα πρόοδου, αποδεικνύουν ότι οι αρνητικές πρακτικές ακόμα παραμένουν. Και πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα θέματα, η όξυνση της κατάστασης, η επίταση αυτών των δυναμένων επηρεάζει όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες και τα παιδιά τους. Ο στόχος είναι οι άνδρες, οι οικογένειες οι ίδιες και οι παραδοσιακές αξίες. Οι παραδοσιακές αξίες είναι πραγματικά ε, επιβλαβή αυτά τα στερεότυπα. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η νοοτροπία, επειδή υπάρχει αυτή η ιδεολογία, ακόμα και άνδρες χάνουν. Και στόχος των ιδεολογικών, των ιδεολογικών αυτών ιδεολογιών αυτών είναι ακριβώ να διχάσει τον κόσμο. Όσοι δεν είναι, από την μας, όσοι είναι μαζί μα, είναι εναντίον μα δηλαδή. Και εδώ έχουμε ε, θέσει πολύ σκληρέ. Ε, κάποιοι όμω πρέπει να αναλάβουν το ρόλο γιατί λέμε ότι οι γυναίκε, οι εκτεβιστέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να υψώσουμε ε, το ανάστημά μα και να υψώσουμε και τη φωνή μα. Είπαμε προηγουμένω ότι είναι τόσα χρόνια από την επέτειο λειτουργία τη Επιτροπή μα. Ναι, μια από τι συμμετέχουσε στην εκδήλωση είπε ότι δεν μπορούμε να σηκωθούμε απλώ και να ψώσουμε τη φωνή μα. Αν δεν μπορούμε να σηκωθούμε όμω, γιατί δεν το επιτρέπει η κατάσταση, πρέπει να σταθούμε και να συμπεριφερθούμε σαν ε, μια άγκυρα, ένα θεμέλιο που θα επιτρέψει να ξεκινήσει ε, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Αυτό που χρειαζόμαστε και μου αρέσει αυτή η γαλλική έκφραση είναι οι άνθρωποι με αξίε σε αυτόν τον αγώνα. Οι άνθρωποι που είναι Ε, εδώ πρέπει να ε, αναλάβουμε έναν ηγετικό ρόλο ε, για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχει κανένα κακό σημείο η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το εκμεταλλεύονται στην όλη προσπάθεια προπαγάνδας για να επιτεθούν κατά της ισότητας των γυναικών, των γυναικείων δικαιωμάτων Πρέπει εδώ λοιπόν κάτι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις υπέροχες συνεισφορές σας στη συζήτησή μας. Έχουμε πολλούς ακόμα αγώνες να διεξάγουμε και πολλά να συζητήσουμε. Αυτό δεν ήταν παρά μόνο το πρώτο πάνελ της ακρόασής μας. Στο επόμενο μέρος θα ακούσουμε για τα μέτρα των κρατών μελών για το θέμα αυτό μπορούν να έρθουν στο Προεδρείο οι συμμετέχουσες στο πάνελ. Η κυρία Κλάσιτσε, την οποία χαιρετώ θερμά, είναι η πρώτη από τις προσκεκλημένες μας για και με αποχαιρετώ και τις προσκεκλημένες μας από τον πρώτο γύρο του πάνελ. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο πάνελ. So, äh, Καλώς, ήρθατε κυρία Κλάσιτσεκ και κυρία Τσοπ Πάγκαν. Η κυρία Κλάσιτσεκ είναι νομική πυρογνώμων και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση των δικαιωμάτων στην Κροατία και τι γίνεται με τα 11 μέσα προσφέρονται για την περίπτωση έμφυλης βίας και παραβίαση των γενικών δικαιωμάτων στην χώρα Παρακαλώ, το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόσκλησή της στην ακρόαση αυτή. Είναι τιμή μου να μοιραστώ τις εμπειρίες και τις απόψεις μου μαζί σας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των νομοθετικών ε, λύσεων, σε ό,τι αφορά τα θύματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κροατία. Ξεκινώντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι σήμερα δεν μιλάω εδώ ως εκπρόσωπος οποιασδήποτε κρατικής αρχής, αλλά ως νομικός εμπειρογνώμων σε ζητήματα πολέμου που εκείνη την εποχή δεν ήμουν συμμετοχή μόνο στη διαδικασία ενός νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τα θύματα σεξουαλικής βίας, αλλά και στην συγγραφή των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα της Κροατίας. Ένα μέλος του κοινοβουλίου, όταν ένα μέλος του Κοινοβουλίου είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή. Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Κροατία είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές για περισσότερα από 20 χρόνια. Υπήρξαν θύματα σεξουαλικής βίας που δεν είχαν λάβει τη δέουσα προσοχή. Η τοπική νομοθεσία δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των θυμάτων και σε πολλές περιπτώσεις ζήτησαν γραπτές μαρτυρίες για τα σεξουαλικά εγκλήματα που είχαν διαβραχθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχαν καν καταγγελθεί τα σεξουαλικά εγκλήματα αυτά, ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο για θύματα. Το 2013 μια ομάδα εργασίας στα πλαίσια του Υπουργείου δημιουργήθηκε με στόχο να βρει ένα επαρκές μοντέλο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Παράλληλα έγιναν διάφορες αξιολογήσεις πάλι στα πλαίσια του Υπουργείου, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία σωστή νομοθεσία. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η νομοθεσία αυτή ήταν κάτι το οποίο είχαμε ανάγκη α, απελπισμένα. Έπρεπε άτομα τα οποία υπέφεραν για περισσότερα από 20 χρόνια να μπορέσουν να βρουν δικαίωση. Και αυτό ήταν μια τεράστια πρόκληση. Ε, λόγω του χρόνου που είχε περάσει σε συνδυασμό με τη συνθήκη ποινικοποίηση δεν υπήρχαν συγκεκριμένα δεδομένα για τα θύματα αυτά. Γυναικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί προσπάθησαν να συγκεντρώσουν τα θύματα σεξουαλικής βίας και να μπορέσουν να μας δώσουν στοιχεία για το τι ήταν πραγματικά σημαντικό για τα θύματα αυτά. Οι διεθνείς πολιτικές που καταπολεμούν τη βία ενάντια στις γυναίκες σε γενικά επίσης ε, ε, ε ήταν κάτι το οποίο λάβαμε υπόψη. Πιο συγκεκριμένα, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, παρόλο που δεν είχε ακόμη επικυρωθεί, αναγνωρίστηκε ως τεράστιο ατού στην δημιουργία της νομοθεσίας αυτής και κάποιες από τις αρχές της σύμβασης αυτής έχουν εφαρμοστεί στο, στην νομοθεσία. Ένας από τους ακρογωνιαίους λήθους ήταν ότι η κοινωνία έπρεπε να αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση και τα θύματα της κακοποίησης αυτής, κυρίως οι γυναίκες, ζούσαν με το τραύμα και την εγκατάλειψη της κοινωνίας. Η πρόκληση βεβαίως ήταν να μπορέσουμε να ορίσουμε και την σεξουαλική κακοποίηση, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη διάσταση της φιλετικής διάκρισης, αλλά και να λάβουμε υπόψη μας τον παράγοντα των εγκλημάτων κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα έπρεπε να θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε όλες τις εγκληματικές πράξεις ενάντια στην σεξουαλική ελευθερία που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κροατία. Επομένως δεν ήταν ε, σχετικό κατά πόσο η σεξουαλική βία διαπράχθη ως μια προσωπική εγκληματική ενέργεια ή στα πλαίσια μιας στρατηγικής του πολέμου. Παρόλο που υπήρχε, αν υπήρχε, αν είχε διαπιστωθεί απλώς σχέση ανάμεσα στο έγκλημα και στην περίοδο του πολέμου, αρκούσε. Ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια σύνδεση ανάμεσα στο δράση και στο θύμα. Τα στοιχεία του δράστη, το φύλλο, η εθνικότητα, δεν είχαν καμία σχέση. Το πιο σημαντικό ήταν α, να συνειδητοποιήσουμε κατά πόσο ο δράστης ποτέ διώχθηκε, γιατί ήταν γνωστό και στις αρχές. Αυτό που έπρεπε να εξασφαλίσουμε ήταν ότι όλα τα θύματα θα μπορούσαν να βρουν στήριξη ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, εθνικότητα, ηλικία, φύλλο κτλ. Στα πλαίσια της διοίκησης θα έπρεπε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία της ταυτότητας του θύματος αλλά και την εμπιστευτικότητα, το απόρριτο όλων των στοιχείων τίποτα στην διαδικασία αυτή δεν γίνεται χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του θύματος. Οι συνεντεύξεις συνήθως γίνονται με ψυχολόγους ένας προς έναν, όπου το θύμα λαμβάνει την ψυχολογική στήριξη, που σημαίνει ότι ένα άτομο εμπιστοσύνη μπορεί να βρίσκεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη θυματοποίηση, υπάρχει πάντοτε ε, απόρριτη συλλογή των δεδομένων και σε γενικές γραμμές δεν, δεν ε, υπάρχει ανάγκη για επιπλέον συνεντεύξεις. Με δεδομένο ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υπάρχει καταγεγραμμένο αρχείο των σεξουαλικών εγκλημάτων, μια ανεξάρτητη αρχή συγκροτήθηκε στο Υπουργείο με στόχο να αξιολογήσει κατά πόσο έλαβε χώρα το σεξουαλικό έγκλημα, έτσι όπως περιγράφεται στην ανάλογη νομοθεσία και τι πέφερε το θύμα. Υπήρχε μια επιτροπή από γιατρούς, από νομικούς, από δικαστές, από ψυχολόγους και άλλους εμπειρογνώμονες. Σε ό,τι αφορά τώρα τις νομικές αποζημιώσεις για τα θύματα σεξουαλικής βίας, η νομοθεσία αυτή προέβλεπε ένα συνολικό, μια συνολική αποζημίωση οικονομική αφενός, κάτι το οποίο ε, συχνά αποδίδεται από τους διαδικαστές, αλλά και μηνιαία επιδόματα. Γυναίκες οι οποίες αναγκάστηκαν να κάνουν έκτρωση ή ε, κατέληξαν σε μια εγκυμοσύνη, έχουν την ε, δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερη οικονομική αποζημίωση. Έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική νομική και υγειονομική βοήθεια. Η ψυχολογική στήριξη προβλέπεται και για τα μέλη της, ε, των οικογενειών των θυμάτων. Τα θύματα έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθελψη, θεραπείες σεξουαλικά μεταδόμενων νοσημάτων. Θέλω τώρα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η οικονομική αποζημίωση είναι τεράστια βοήθεια για τα θύματα αυτή, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι το βασικό ζητούμενο που έπρεπε να στο οποίο έπρεπε να επικεντρωθούμε. Ήταν ανάγκη να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το τραύμα για να μπορέσουν να προχωρήσουν τη ζωή τους παρακάτω τα θύματα αυτά. Μιλάω στο να πρέπει να καταφέρουν να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς να επικεντρώνονται σε αυτό το τραύμα διαρκώς, να μπορέσουν να κοιτάξουν προς το μέλλον αντί να επιμένουν στο παρελθόν, να μπορέσουν να επιβιώσουν του τραύματος αυτού. Επομένως, είναι ιδιαίτερα αναγκαία η ψυχολογική στήριξη, η ψυχολογική α, θεραπεία. Και δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο αυτή ήταν επαρκής. Τα θύματα χρειάζεται, χρειάζεται από εμά να αναγνωρίσουμε ότι υπέστησαν σεξουαλική βία και ότι δεν ήταν δική τους ευθύνη. Είναι ανάγκη να υπάρξει μια ανοιχτόμυαλη κοινωνία που να τους προσφέρει την στήριξη που χρειάζονται και να τους επιβεβαιώσει η κάθε κοινότητά τους ότι τα θύματα δεν είναι μόνα τους και η κοινωνία τα αποδέχεται. Η ορθή εφαρμογή Τη νομοθεσία αυτή θα έχει τεράστια ωφέλη όχι μόνο για τα θύματα σεξουαλική βία του πολέμου αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό τη. Είναι σημαντική για την καταπολέμηση των συνεπειών του πολέμου, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα παρόν στη χώρα μα. Αλλά η οθέτηση τη νομοθεσία αυτή στέλνει ένα μήνυμα. Η σεξουαλική βία ενάντια στις γυναίκες δεν θα γίνεται ανεκτή, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Όλα τα θύματα αξίζουν υποστήριξη και προστασία υπάρχει ακόμη ένας τεράστιο αριθμός θυμάτων που ζουν στη σιωπή και που δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στο σύστημα. Επομένως, στόχος της νομοθεσία αυτής είναι, θα έχει εκπληρωθεί μάλλον, όταν όλα η πλειοψηφία των θυμάτων αυτών έχουν καταφέρει να επιτύχουν αυτό το οποίο έχουν ανάγκη. Περισσότερα θύματα έρχονται, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις αρχές, ώστε να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα δεδομένων έναντι συμπεράσματος. Δεν υπάρχει τέλεια νομοθεσία. Η εφαρμογή του νόμου αυτού και η αξιολόγηση του θα δείξει πόσο επωφελής ήταν και τι πρέπει να κάνουμε ακόμα. Να σας πω απλώς ότι για την Κροατία χρειάστηκαν 20 χρόνια για να αναγνωρίσει το γεγονός ότι η σεξουαλική βία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Η λύση του προβλήματος αυτού προέκυψε από την ανάγκη των θυμάτων και η Κροατία βρήκε τη δύναμη να αναγνωρίσει το λάθος και να το αντιμετωπίσει. Με δικά της μέσα η χώρα χρησιμοποίησε τοπικούς εμπειρογνώμονες, εφάρμοσε διεθνή στάνταρ και μια συγκεκριμένη νομοθεσία που προβλέπει η συνολική προστασία των θυμάτων. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι απλώς μέρος της λύσης του προβλήματος. Η αξιολόγηση θα μπορέσει να δείξει κατά πόσο εμείς αποδώσαμε δικαιοσύνη στα θύματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην ξεπέρασα το χρόνο μου. Πολύ σας ευχαριστούμε για αυτές τις διαφωτιστικές πληροφορίες, γιατί είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για, όλη, για τον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τώρα η τελευταία μας ε, προσκεκλημένη για αυτό το πάνελ, η κυρία Τσόπ Πάγκαν, για το επόμενο κύμα σε σχέση με την ε, βία, ε, την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και το τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν ε, από την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στα κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν θα πάρετε το λόγο για 15 λεπτά και να συγχωρείτε Δεν το ήξερα, κυρία Τσοπάγκαν. Να σας δώσω το λόγο, διότι έχουμε επιπλέον 15 λεπτά τους διερμηνείς μας. Οπότε μετά θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε και μια σύντομη παρουσίαση από την ΕΙΚΕ, από το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Οπότε Πραγματικά λυπούμε που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο. Ήταν συναρπαστικέ οι παρουσιάσει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Οπότε τώρα ε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχετε τον λόγο, κυρία Τσόπ Πάγκαν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω καλά το χρόνο μου. Πρώτα απ' όλα για την WAVE, την οργάνωσή μας. Είμαστε ένα δίκτυο 153 οργανώσεων γυναικών. Εκπροσωπούμε 46 χώρες της Ένωσης και εκτός Ένωσης. Δημιουργηθήκαμε για, λόγω της ανάγκης υπεράσπισης των, των δικαιωμάτων των γυναικών. Είμαστε μια συλλογική φωνή. Οι πληροφορίες ε, που δίνουμε είναι πολύτιμες, προέρχονται από το τι συμβαίνει ε, στην κοινωνία και βεβαίως χρειάζεται αυτό στο δικό σας επίπεδο. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ. Δυστυχώς, όπως ελέγχθη νωρίτερα από τους προηγούμενους ομιλητές, υπάρχουν πολύ έντονα κινήματα κατά των γυναικών. Έχουν αντικοποιήσει τη δράση τους, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Όπως είπα νωρίτερα, αυτά τα ακροδεξιά κινήματα προωθούν μεταρρυθμίσεις νομοθετικές που ε, πλήττουν τις γυναίκες, ε, που πλήττουν τις οργανώσεις των γυναικών ε, και επίσης στρεβλώνουν το μήνυμα των φεμινιστικών οργανώσεων. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει σε ό,τι αφορά τη σύμβαση για να μπορούν οι γονείς να υιοθετούν παιδιά, ε, πρέπει να υπάρχει καλή θέληση ε, για την συνεργασία με το παιδί και υπάρχει το θέμα της κυδαιμονίας ε, του παιδιού ε, δεν δημιουργούμε ασφαλές περιβάλλον ε, για τα παιδιά αυτά. Επίσης αυτοί που έχουν προβεί ε, σε καταχρήσεις ε, έχουν τον τρόπο να συνεχίσουν να προβαίνουν στις καταχρήσεις αυτές. Δίνουν μάχες και δικαστικά. Μια ομάδα πυρογνωμόνων τέλη Μαρτίου εξέδωσε μια δήλωση για την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό της βίας κατά των γυναικών και μάλλον σε ό,τι αφορά την, την κυδαιμονία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γυναίκε έχουν δικαίωμα ιδιαίτερη υποστήριξης, τα παιδιά έχουν δικαίωμα ιδιαίτερη υποστήριξη, όπω και οι γυναίκε. Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι επιπτώσει είναι δραματικέ ε, τη ενδοκινιακή βία για τα παιδιά. Ε, και αυτό βεβαίω έχει επιρροή και στι επόμενε γενναίε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ε, όλη τη στρατηγική και δουλειά ανάπτυξη για να δούμε τα πράγματα από την προοπτική των παιδιών είναι κάτι το οποίο αγνοείται από τις ομάδες αυτές. Ε, ακούγονται και κάτι επιχειρήματα τα οποία είναι απίστευτα, ότι το παιδί πρέπει ούτως ή άλλως κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει την κατάχρηση των παιδιών, γιατί να μην συμβεί το, τον, ε, τώρα, ό,τι αργότερα. Σε ό,τι αφορά που είναι σε ανάγκη στο άρθρο 1, ε, λέγεται στη σχετική οδηγία τα, τα, τα θύματα του εγκλήματο πρέπει να τύχουν επαγγελματική και ευαίσθητη μεταχείρισης, Λαμβάνοντα υπόψη τις ιδιαίτερε ανάγκες των θυμάτων. Έχουμε πληροφορίες ότι 44% των θυμάτων θεωρούν ότι η διαδικασία μάλλον τους έκανε μεγαλύτερη ζημιά από τη, τη ζημιά που τους, που τους προκάλεσε ο δράστης. Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος για να μην κατηγορούνται τα θύματα επειδή είναι θύματα και να μην έχουμε μια δεύτερη τραυματική εμπειρία. Είναι σημαντική η κατάρτιση των επαγγελματιών, αλλά δεν αρκεί. Επίσης, όλο και πιο συχνά γίνεται μια δουλειά σε επίπεδο επικοινωνίες ε, με τους δράστες Το βασικό ζήτημα όμως τώρα, όταν έχουμε ένα βιασμό ή ενδοκρινική βία, είναι ποιος βοηθάει τελικά τους δράστες. Γίνονται και φιλοσοφικές συζητήσεις στα δικαστήρια την περσμένη εβδομάδα. Ένας δικαστής, ε, στη δικαρτία και της ακρόασης, λέμε ότι μια γυναίκα δέχεται ενίσχυση από κέντρα γυναικών, ενώ ένα άντρα δεν έχει κάτι αντίστοιχο και ότι αυτό αποτελεί διάκριση. Πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν την ισότητα. Αυτό που μπορεί να κάνει η Επιτροπή Γυναικών είναι να ζητήσει να υπάρχουν μηχανισμοί που θα εξασφαλίζουν ότι οι χώρες θα λαμβάνουν υπόψη αυτές την κακοποίηση κάθε φορά. Έχει υποθεί και από υπηρεσίες υποστήριξης γυναικών και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, για την κυδαιμονία ότι υπάρχουν απαιτήσει έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βία του συντρόφου. Αυτό υποτίθεται ισχύει στη θεωρία, στην πράξη δεν ισχύει πρέπει να γίνει σαφές ότι όλοι οι δράστες ε, ε πρέπει και αυτοί να λαμβάνουν βοήθεια, αλλά δεν πρέπει τα χρήματα αυτά να προέρχονται από τα χρήματα που λαμβάνουν οι γυναίκες, διότι έτσι θα, μειωθεί η χρηματοδότηση. Υπάρχουν ε, οι γραμμές ε, τηλεφωνικές, υπάρχουν τα καταλήμματα. Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί η διετής έκθεσή μας ε, και βεβαίως η Επιτροπή ΦΕΜ θα λάβει τις πληροφορίες μόλις υπάρξουν. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά λείπουν χιλιάδες καταλήμματα παρότι η διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης το προβλέπει. Μόλις 40% των ευρωπαϊκών χωρών της Ένωσης έχουν ένα κρεβάτι, ένα κατάλημα ανά 100.000 κατοίκου, ανά 10.000 κατοίκου, όπω προβλέπεται από τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Επίση, συχνά χρησιμοποιούνται χρήματα τη Ένωση ε, για την ε, χρηματοδότηση ε, καταλημάτων και χώρων στέγασης, αλλά υπάρχουν και περιοριστικοί όροι για αυτή τη χρηματοδότηση. Έχουμε διαπιστώσει ότι όταν πιέζουμε να υπάρχει να υπάρχει ουδετερότητα ε, σε επίπεδο φύλου. Ε, τελικά υπάρχει λιγότερη χρηματοδότηση από ό,τι στο παρελθόν για τις γυναίκες, διότι υπάρχουν κέντρα τα οποία αφορούν αποκλειστικά γυναίκες και παιδιά. Κάποια παραδείγματα ε, ε, του κινήματος κατά των γυναικών. Τον Αύγουστο κάποιος μας είπε ότι η ΜΚΟ της Τσεχίας σε μία ακρόαση υπόθηκε ότι η χρηματοδότηση που υπήρχε από το 2016 δεν εγκρίθηκε και πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα. Διότι τα χρήματα προχώρησαν από τα μία ταμεία της Ένωσης και δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ε, για τέτοιου είδου ε, συμβουλές. Ε, μάλλον ε, νομική βοήθεια για τις γυναίκες. Ε, χρησιμοποιείται λοιπόν αυτό Ω ε, δικαιολογία για να μην υπάρχει καμία ασφάλεια για τι γυναίκε. Έχουμε παραδείγματα από πολλέ χώρε. και από τι 46 χώρε. και ανάλογα με το ποια χώρα σα ενδιαφέρει μπορούμε να σα δώσουμε στα στοιχεία αυτά. Να μα τα ζητήσετε, παρακαλώ. Αυτό που μπορεί να κάνει η ΦΕΜ είναι να πιέζει ε, για κοινά πρότυπα τα οποία θα σέβονται όλε οι χώρε και τα νέα κράτη-μέλη. Εμεί ω ΜΚΟ προσπαθούμε, ε, προσπαθούμε να του κάνουμε να λογοδοτήσουν και στις χώρες μας ε, δεν μας αγαπούν ιδιαίτερα. Χρειαζόμαστε βοήθεια, λοιπόν, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την συναρπαστική παρουσίαση και τώρα ο κύριος Μάτιτς έχει ζητήσει το λόγο και μετά η κυρία Ραφαήλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σήμερα είναι θλιβερή επέτειος της κατάληψης της πόλης μου στην Κροατία στο Βούκοβάρο που όταν εισέβαλαν οι Σερβοί ε, δολοφονήθηκαν άνδρες και γυναίκες, βιάστηκαν, θανατώθηκαν. Πολλοί από εμά πήγαμε σε τρόπο συγκέντρωση σε όλη τη Σερβία. Και εγώ βεβαίω υπήρξα μάρτυρα αυτών των γεγονότων. 20 χρόνια αργότερα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα. Στην δική μου σοσιαλιστική ε, κυβέρνηση είχα την τύχη να γίνω υπουργό των βετεράνων για το θέμα αυτό και αποφάσισα να προβλεφθεί αποζημίωση για τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων στους καιρούς του πολέμου. Ήταν πολύ δύσκολο να πετύχει αυτό, γιατί ξέρετε ότι σε κανονικές συνθήκες πρέπει να υπάρξει και το θύμα και ο δράστης και να κρυθούν. Στα 20 χρόνια όμως αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ατιμορρησία και καμία δικαιοσύνη για τα θύματα. Αποφασίσαμε λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση και να αλλάξει και ο νόμος. Και το πετύχαμε. Είναι ο, προ, ο μόνος τέτοιος νόμος ε, στην πρώην, ε, δημοκρα... στην πρώην Ιουκοσλαβία, αλλά είναι και ο μόνος στην Ευρώπη, δυστυχώς. Χρειαζόταν, γιατί τα θύματα Ε, χρειαζόταν γιατί έτσι τα θύματα μόνο μία φορά αναγκάζονται να προσέλθουν στους δικαστές και στους ιατρικούς, στους ιατρούς ανακριτές που διαπιστώνουν την περίπτωσή τους. Αποφασίσαμε λοιπόν να τις υποστηρίξουμε και οικονομικά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η υπόθεση μπορεί να συνεχιστεί στην εκδίκασή της, απλώς μετά τον πόλεμο είναι πολύ δύσκολο να δοθεί συνέχεια, γιατί έχει μεσολαβεί, έχω μεσολαβεί τέτοια γεγονότα που το μόνο που μπορεί να ξέρει το θέμα είναι ότι ήταν Σέρβος. Και ε, πραγματικά με τα στοιχεία που έχω και την εμπειρία που αποκτήσαμε από τα γεγονότα αυτά, ευχαριστώ να δώσω πληροφορίε και σε όποιον συνάδελφο τη επιθυμεί. Ευχαριστούμε. Θερμέ ευχαριστίε. Σαμίρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για, την παρουσία, για τις παρουσίες σας και το εκτιμώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πιστήσω την προσοχή σα στο γεγονός ότι υπάρχει ένα θέμα διαφυλετικό της εμφυλής ε, κατά των γυναικών δηλαδή. Βάσει του, του λόμπι για τις γυναίκες ε, στην Ευρώπη, οι γυναίκες... 30% ε, γυναικών χωρί χαρτιά έχουν υποστεί ω μετανάστριε βία την τελευταία χρονιά και 40% γυναικών με ειδικέ ανάγκε έχουν περισσότερε πιθανότητε να υποστούν ε, βία. Είναι πιο δύσκολο λοιπόν να βρούμε κέντρα υποστήριξη όπου μπορούν να καταφύγουν οι γυναίκε αυτέ. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα και η ερώτησή μου είναι, ξέρετε, ποιε είναι οι καλύτερε πρακτικέ στα κάτι που σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν τι ανάγκε τέτοιων συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων γυναικών και πώ μπορούν τα κατημέλη αλλά και μη κυβερνητικέ οργανώσει να, να λάβουν συγκεκριμένη δράση για να βοηθήσουν αυτές τις γυναίκες και να, μπορέσει, ε, να μπορέσουν να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να έχουν πρόσβαση σε κάποιο κέντρο υποστηρίξης για τις γυναίκες χωρίς ε, ε, νόμιμα έγγραφα. Πώς θα μπορέσουν οι καταγγελίες τους για βία να ληφθούν υπόψη σοβαρά από τα κάτι μελη και να μην συνεχίσουν να μένουν εκτεθειμένες. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με την βία στο διαδίκτυο. 9 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια είναι διαρκώς εκτεθειμένα, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Ε, ποια η άποψή σας για την ευρωπαϊκή οδηγία που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα τη βία κατά των γυναικών και τις επιγραμμικές προεκτάσεις της. Ευχαριστούμε. Jackie Jones και μετά ο κύριος Μπρένερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κάθε μια από εσά για τις παρουσιάσεις σας και εσάς συνάδελφε να ρωτήσω για τα διαφορετικά ταμεία. Μπορείτε να πείτε περισσότερα στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Γυναικών. Βέβαια τώρα δεν έχουμε χρόνο, αλλά θα μπορούσατε να μας στείλατε περισσότερες λεπτομέρειες στοιχεία για το αν τα κονδύλια αυτά έχουν ε, υπάρξει για τα κονδύλια μάλλον αυτά έχουν υπάρξει περιπτώσει κακοδιαχείριση στα κράτη-μέλη. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Ευχαριστούμε, κυρία Μπρένε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια αντίδραση για να πω ότι η νομοθεσία του κάθε τους μέλους δυστυχώς ε, δεν είναι αρκετή. Είχαμε μια πρόσφατη υπόθεση στην Γαλλία. Υπάρχει πλημέλημα στην ε, ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων και η αστυνομική και δικαστική ε, καλή βούληση ε, δεν αρκεί για την πρόβλεψη ασφαλιστικών μέτρων σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιταχύνουμε και να επιτείνουμε την δράση μας. Δεν μπορούμε να ε, ξεχνάμε τις περιπτώσεις εζυγικής βίας και να το συγχωρούμε αυτό λόγω του θρησκευτικού, των θρησκευτικών επιθύσεων του θρησκεύματο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κλάσιτσεκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί δεν έχουμε χρόνο. Το βασικό ζήτημα στη Κροατία, εφόσον αναφερόμαστε σε θύματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν υπάρχουν πολλά κράτη που να έχουν μια πρόσφατη ανάλογη εμπειρία. Επομένως, η νομοθεσία αυτή ήταν, τολμώ να πω, μοναδική. Γιατί δεν είχαμε κάποιο παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Αυτό που κάναμε ήταν να συλλέξουμε πολλές πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η αξιολόγηση του νόμου αυτού θα δείξει κατά πόσο επιτύχαμε. Ελπίζω γιατί πάντοτε υπάρχει χώρος για βελτίωση. Τα δεδομένα είναι ένα σημαντικό ζήτημα για μας, παραμένει, γιατί δεν υπάρχει η εκτίμηση εκείνη την εποχή όταν προσπαθήσαμε, προσπαθούσαμε να συστήσουμε την νομοθεσία εκτιμούσαμε ότι υπάρχουν χιλιάδες θύματα, αλλά μόλις ε, μερικές εκατοντάδες ήρθαν σε μας. Όπως είπα λοιπόν, είναι ανάγκη να προωθήσουμε τον νόμο αυτό, το ώστε να έχουμε περισσότερα δεδομένα και να έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Αυτό παραμένει ένα βασικό πρόβλημα στην Κροατία. Πώς μπορούν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί να, να επωφεληθούν; πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ακριβώ αυτοί οι οργανισμοί έρχονται σε επαφή, μάλλον πώς μπορούν να μας βοηθήσουν. Αυτοί είναι που έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα, επομένως ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός και η δουλειά τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μας. Νομίζω ότι υπήρξε και ένα ερώτημα σχετικά με το πώς οι αρχές, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αρχές παίρνουν τα θύματα αυτά σοβαρά να σας πω ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που μπορούμε να λάβουμε προς αυτό το σκοπό. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς ήταν η εκπαίδευση των επαγγελματιών. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν και αυτό το οποίο κάναμε. Από και πριν α, θέσουμε σε εφαρμογή την νομοθεσία, είχαμε αρκετά προγράμματα κατάρτισης για τις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα θύματα, να μπορέσουν να καταλάβουν το επίπεδο βίας που είχε συντελεστεί, να βοηθήσουν τα θύματα να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Δεν είμαι σίγουρη στο κατά πόσο σας απάντησα. Αυτά έχω να πω εγώ από μεριά μου. Ναι, να προσθέσω κάτι το θέμα των εθνικών ταμείων είναι καλύτερο να προχωρήσουμε έτσι. Πρέπει να ορίσουμε πληροφορίε έτσι κι αλλιώ. Οι γυναίκε με αναπηρία, οι γυναίκε χωρί χαρτιά. Ναι, βεβαίω, τεράστιο ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι μια γυναίκα χωρί χαρτιά από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ΜΚΟ που βοηθούν θύματα τότε ναι υπάρχει βοήθεια όταν όμως ε, πέφτουν στα χέρια του κράτους τα θύματα ε, θα πρέπει να δώσουν τα ονόματά τους, θα πρέπει να καταγραφούν. Και δεν είναι καλό για αυτούς. Ε, είναι και κίνδυνο θα έλεγα. Ε, γι' αυτό λοιπόν εδώ πάλι στηρίζουμε αυτό που λέει η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, ότι η ΜΚΟ πρέπει να είναι ένας κεντρικός παράγοντας που θα παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Οι γυναίκες με αναπηρία, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν έχουμε ακόμα αρκετές υπηρεσίες ε, στέγασης ε, για αυτές τις γυναίκες. Ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετωπίσης του θέματο. Προσπαθούμε να έρθουμε όσο γίνεται πιο κοντά στι γυναίκε διότι τα φόρουμ μάλλον οι μορφές αναπηρίας είναι πολλές και διάφορες είναι δύσκολο να βρεθεί ένας τόπος διαμονής ο οποίος να ταιριάζει σε όλους έτσι λοιπόν η νομοθεσία που μας επιτρέπει να απομακρύνουμε το δράστη από το σπίτι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες με αναπηρία που, είναι, που έχουν υποχθεί σε βία για να μπορούν να μείνουν στο δικό τους περιβάλλον. Ζητούμε λοιπόν από τις ε, οργανώσεις ε, ε, να μπορούν εκεί να πάνε και να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Βεβαίως υπάρχουν διάφορα επίπεδα, διάφορα που μπορούν να γίνουν, αλλά δεν είναι πάντα ασφαλή, ασφαλής αυτές οι λύσεις. Αυτά, για να μην κλέψω και χρόνο άλλων. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες σας, σε όλες τις εμπειρογνώμονες σήμερα και τους βουλευτές και τις βουλευτές για το πάθος με το οποίο έκαναν τις παρεμβάσεις τους και την πειθαρχία. Ε, όλες ε, παρουσιάσεις δυστυχώς υποβλήθηκαν στον κανόνα αυτή της πειθαρχία, αλλά έχουμε πραγματικά ε, αρκετά που δεν έχουν κυρώσει τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης οπότε καλό είναι να παρουσιάσετε και εσείς με τη σειρά σας τα υπόθηκαν εδώ στους αρμόδιους για να κάνουν κάτι και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία όλοι μεταξύ μας να εμβαθύνουμε κάπως στην γνωριμία και στο κοκτέιλ που θα πιούμε όλοι μαζί και να ε, συνεχίσουμε τη συζήτησή μα. Είμαστε σχεδόν στο τέλος τη συνεδρίαση, αλλά δεν θέλω να αφήσουμε την ε, παρουσίαση από την ε, προκεκλημένη μας από το ΙΓΕ. Η κυρία Πετσιουρένε. Παρακαλώ μια πολύ σύντομη παρουσίαση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα στην ε, πρακτική ε, ζωή, γιατί έχετε ετοιμάσει αυτό τον ε, οδηγό για τις αστυνομικές αρχές για την περίπτωση της ενδοικογενειακής βίας κατά των γυναικών. Έχετε κάνει φοβερή δουλειά και νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί και εδώ αυτό. Έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο για να σας ακούσουμε. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής ΦΑΜ, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τόσα κάνουμε με την αξιολόγηση κινδύνου και την αξιολόγηση επιπτώσεων. Εδώ λοιπόν μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με τη, με τη διάσταση της υλοποίησης. Μου ζητήθηκε να είμαι πολύ σύντομη και Ξέρω ότι και εσείς μπορείτε να προωθήσετε και να υποστηρίξετε τις ε, κατευθύνες γραμμές που εκπονήσαμε και που είναι διαθέσιμες και εδώ. Οι αριθμοί βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς εμφανίζονται τέτοια κρούσματα, είναι όλα αυτά παράδεκτα οι αριθμοί που βλέπουμε. Ε, η Βίγαν των γυναικών από τους κοντινούς τους, ε, κυρίως συντρόφους και συζύγους, είναι πρόβλημα όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για και την κοινωνία, γιατί το οικονομικό κόστος έχει πολύ αρνητικό, τριπλό αντίκτυπο και στους ίδιους τους άντρες και στο δημόσιο και κοινωνικό μας βίο. Για τις περισσότερες γυναίκες που γνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις βίας, το πρώτο σημείο που απευθύνονται είναι η αστυνομία. Και η αστυνομία μπορεί να επιτρέψει να αποφευχθούν σε κάποιε περιπτώσει οι επανειλημμένε κοινέ βίε, τα κρούσματα βία και των γυναικών ή των παιδιών, εφόσον καταγγελία γίνει ε, γέρο. Και ε, έτσι αυτό, εφόσον υπάρχει σωστή αντίδραση από την αστυνομία, ενισχύει και την εμπιστοσύνη προ τι διοικητικέ αρχέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κοιτάξει τη βία γενικότερα και την ε, υποχρέωση να προστατεύει από την δευτερογενή θυματοποίηση, για να το πω έτσι και πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα μέτρα που έρχονται από την αξιολόγηση κινδύνου και το πώ μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το σύστημα αυτό. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τι περιπτώσει επανειλημμένων κρουσμάτων βία, έχοντα υπόψη τη, τα μέτρα αξιολόγηση του κινδύνου, πράγματα που είναι καθοριστικοί παράμετροι και τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Μα ενδιαφέρει πώ θα εφαρμοστούν σωστά οι νομικέ υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη και για να ε, μεγιστοποιηθεί το επίπεδο προστασία των θυμάτων θα πρέπει να δούμε τη διαχείριση των κινδύνων μαζί με όλου του άλλους όταν σχεδιάζονται παρεμβάσει για τα θύματα. Προστιγμένη διαχείριση του κινδύνου δεν λαμβάνεται επαρκώ υπόψη. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας, αλλά δυστυχώς η Γερμανία πρέπει να διακοπεί στο προβλεπόμενο χρόνο ολόκληρης της συνεδρίασης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Partner violence and allows to estimate accurately the risk that we are facing. Through this, it reduces the threat posed by the perpetrator and protects victims and their children from repeated violence. Risk management